Colleagues, good afternoon. Λοιπόν, γεια σας. Συνάδελφοι, καλώς και πάλι για το δεύτερο ήμιση της σημερινής τόσο ενδιαφέρουσας ημέρας. Έχουμε τώρα την πρώτη ακρόαση του απογεύματος. Καλωσορίζω θερμότατα τον καθηγητή κύριο Μπόρχεστ, όπως Ολλανδικά προφέρεται. Ωραία, μπράβο. Προφέσορ Κάι Μπόρχεστ, καθηγητής ηλεκτρονικών συστημάτων αυτοκινήτων στο Πανεπιστήμιο του Ασάφενμπουργκ. Είναι Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών. Άσεμπερς λέει, έτσι λέει, προφέρεται στην τόπια διάλεκτο. Μάλιστα. Έχετε ε, εσείς ε, συστήσει αυτό το κέντρο και το πρόγραμμα το αντίστοιχο και χωρίς καμιά αμφιβολία είστε ο άνθρωπός μας ο ειδικό που ψάχναμε. Σας δίνω το λόγο για 10 λεπτά, παρακαλώ πολύ. Θα προσπαθήσω να σας εξεπλήσω σε 10 λεπτά αυτό που εξηγώ σε 90 λεπτά στους φοιτητές μου. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε τα πιο βασικά ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στο 10 λεπτό. Θα σας δώσω ποιες είναι οι ουσίες οι οποίες μολύνουν από τους κινητήρες πετρελαίου, πώς δημιουργούνται και τι μπορούμε να κάνουμε αφού δημιουργηθούν, τα αντίμετρα. Κάποιες ε, μορφές προστασίας, πρόληψης, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο όχι πολυτίμιο από ορισμένου όπως ξέρουμε, είναι η λεγόμενη προστασία του κινητήρα να δούμε πόσο ε, υποχρεωτικό και χρήσιμο είναι αυτό και τι δυνατότητες υπάρχουν για τεχνικές ε, βελτίωσεις. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες δυνατότητες αλλά δυστυχώς κοστίζουν. Βλέπουμε εδώ κάποιες από τις ουσίες αυτές οι οποίες προέρχονται από τις μηχανές ε, εσωτερικής καύσης και ιδιαίτερα τις πετρελαιο, τους πετρελαιοκινητήρους. Βλέπετε εσείς τα τυπικά προβλήματα είναι η εθάλη ή καπνιά, όπως και τα PAH τα οποία ε, ε, ε, δημιουργούν, είναι καρκινογόνα. Το αντίμετρο είναι γνωστό, είναι να να εγκαθιστούμε ένα φίλτρο συλλογή σωματιδίων. Δεν είναι τέλειος ο μηχανισμός αυτός, αλλά μέχρι τώρα είναι μια λύση. Έχουμε όμως βασικό πρόβλημα με τα οξύδια του αζότου. Υπάρχουν δύο είδη οξυδίων του αζότου, το NO και το NO2. Το NO είναι ασταθές στην ατμόσφαιρα και οξυδώνεται ε, ταχύτατα, ενώ το NO2 παραμένει, μυρίζει άσχημα, δημιουργεί πρόβλημα στο αναπνευστικό, είναι υπεύθυνο για την τοξική βροχή, για την, για την όξινη βροχή ε, για το πρόβλημα του ε, καταλυτικού λεγόμενου όζοντος, όπως επίσης και για το PNA. Και ε, δημιουργεί και αυτό, υπάρχουν υποψίες για καρκίνο, ενώ προκαλεί ερεθισμό του αναπνευστικού και τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν ξεπερνούν τα ανεκτά επίπεδα εκπομπής NO2. Περνάμε στην επόμενη αν θέλετε τώρα διαφάνεια. Πώς μπορούμε εμείς να μαζέψουμε αυτές τις ουσίες. Αν το κάνουμε με τέλειο τρόπο παίρνουμε μόνο μετά την καύση ε, διοξίδιο του άνθρακα και νερό, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό και έχουμε διαφορετικές επιπλέον ουσίες πλέον του διοξιδίου και του νερού. Σε επίπεδο σωματιδίων έχουμε να κάνουμε με το μονοξίδιο του αζότου όπως επίσης και το μονοξίδιο του ε, άνθρακα. Εάν λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία ο κινητήρας και δεν είναι επαρκής ο κύκλος της καύσης, ενώ αντίθετα δημιουργείται διοξίδιο του άνθρακα. Ενώ από την άλλη αν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της καύσης, τότε έχουμε εκπομπή ακριβώς διοξιδίου του αζότου. Έχουμε λοιπόν δύο αντιφατικούς στόχους. Από τη μία υψηλή εθερμοκρασία αυξάνει την αποδοτικότητα του πετρελαιοκινητήρα, καίει την καπνιά, την εθάλη, δεν θα έχουμε πρόβλημα εθάλης, αλλά θα δημιουργεί πάρα πολλές ποσότητες διοξιδίου του αζότου. Αν ο πετρελαιοκινητήρας δουλεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες, δημιουργείται εθάλη, η ισχύ της μηχανής μειώνεται, η αποδοτικότητα επίσης, αλλά δεν εκπέμπουμε διοξίδιο του αζότου. Έχουμε λοιπόν μια δύσκολη επιλογή να κάνουμε όταν σταθμίζουμε το σωστό επίπεδο λειτουργίας της μηχανής και το λογισμικό που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει παραμέτρους που επιτρέπουν στους κατασκευαστές να βρουνε μια βέλτιστη συμβιβαστική όμως πρόταση. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό. Αυτό είναι βασικά πως ε, δουλεύει ο αέρας μέσα στον κινητήρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μετρονόμο αέρα θα λέγαμε που υπολογίζει ακριβώς ε, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τις ποσότητες. Υπάρχει ο πολλαπλασιαστής ουσιαστικά ισχύος ο οποίος χρησιμοποιείται τώρα κυρίως και το πιο σημαντικό εδώ είναι η κυκλοφορία των αερίων της εξάτμισης. Βλέπετε εδώ στον πίνακα ότι περνούν μέσα από μια βαλβίδα εξόδου που ελέγχεται και αυτή και ανακατεύεται με τον φρέσκο αέρα τον οποίο καταπίνει ο κινητήρας και αυτό βοηθά να κατεβαίνουν οι πολύ ψηλέ θερμοκρασίες της καύσης. Έχουμε και κάποια επιπλέον στοιχεία εδώ. Χρησιμοποιούμε επίσης και τον, τη βαλβίδα EGR για τον έλεγχο πάλι της κυκλοφορίας του αέρα και πολύ συχνά έχουμε και ένα βοηθητικό πολλαπλασιαστή ισχύω το intercooler που χρησιμοποιεί εκ νέου τα αέρια της εξάτμισης σε χαμηλές θερμοκρασίες για την αύξηση της ισχύω της μηχανής, κάτι το οποίο όμως δυστυχώς κατεβάζει την θερμοκρασία της καύσης για μια ακόμη φορά. Ένα άλλο αντίμετρο είναι το, η επιλεκτική καταλυτική μείωση. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται συμπληρωματικά. Αυτό που βλέπετε εδώ λοιπόν είναι στην ουσία ένα χημικό εργοστάσιο μέσα στο, στο, στο τμήμα που είναι η μηχανή. Αυτό το SCR περιλαμβάνει ένα ειδικό καταλήτη. Υπάρχει ε, ένα διάλειμμα ουρίας το οποίο εγχέεται ε, μαζί με αμμονία και αυτά όλα ε, επηρεάζουν την εκπομπή μονοξιδίου του αζότου και βγαίνουν και τα υπόλοιπα συστατικά εφόσον όλα βέβαια δουλεύουν σωστά. Αυτό το σχήμα είναι υπεραπλουστευμένο βέβαια. Υπάρχουν ε, και άλλα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η επελεκτική καταλυτική μείωση. Η τεχνολογία αυτή είναι επιτυχής εδώ και χρόνια για τα φορτηγά. Δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ για τα γιοταχή ε, ίσως να χρησιμοποιείται περισσότερο στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου οι απαιτήσει επίπεδο εκπομπών είναι αυστερότερες. Υπάρχει επίσης ένας άλλος καταλήτης ο οποίος είναι φινότερος αλλά λιγότερο αποτελεσματικός, ο LMT ο οποίος μαζεύει με χημικό τρόπο το άζωτο, συλλαμβάνεται λοιπόν η ποσότητα αυτή και στην ουσία ε, γίνεται μια εκ νέου επεξεργασία και ανάμιξη με ένα ιδιαίτερα πλούσιο μείγμα και αποσυντίθεται με το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι ένα πολύ περίπλοκο σύστημα αλλά και αυτό δουλεύει αρκετά καλά. Ο έλεγχος των συστημάτων μπορεί να γίνεται από μία μονάδα ελέγχου αυτόνομη ή να αποτελεί τμήμα του συστήματος της μονάδας ελέγχου του συνόλου του αυτοκινήτου ή να συνεργάζονται οι δύο αυτές μονάδες ελέγχου στενά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην πράξη ποιο είναι, ότι είναι πολύ χαμηλές οι, ε, θερμοκρασίες και ε, έχουμε συγκέντρωση νερού και εθάλης καπνιάς και ε, αυτό τι σημαίνει στο ECR ότι είναι πολύ μεγάλη η ε, θερμοκρασία και εκλείεται αμμονία από τον καταλήτη και επίσης αν οι ακραίες θερμοκρασίες περιορίζεται η λειτουργία. Μπορεί να υπάρχει ένας περιορισμός Και αν είμαστε σε αυτό το κύκλο είναι πολύ ε, ύποπτο να χρησιμοποιείτε μια συσκευή που περιορίζει τη δυνατότητα αυτή. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες διάφορες να βελτιωθούν αυτές οι λειτουργίες και να διαβρεθεί αυτή η θηρίδα ε, θερμοκρασιών. Σας τα αναφέρω εδώ, υπάρχουν κάποια τεχνικά μέτρα, αλλά αυτό μπορεί ε, να συνάδει με κάποιες θηρίδες ε, θερμοκρασίας και περισσότερο από 17 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα ε, κοστίζουν. Ορισμένα είναι σχετικά συγκρατημένου κόστους, αλλά ε, το εσωτερικό EGR είναι παράκριβο και φυσικά ο κατασκευαστής, αν δεν πιεστεί, θα διαλέξει την πιο φθηνή λύση. Μερικά μέτρα βοηθούν ας πούμε κάποια υλικά που αθίστανται στις θερμοκρασίες, ε, ειδικοί τύποι καταλυτών ε, που αντέχουν σε διάφορες θερμοκρασίες. Αυτό εξαρτάται από τους υπολογισμούς κάθε φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και μπορούμε να περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Ελπίζω να τα καταλάβατε όλοι. Λοιπόν, αρχίζουμε από τους ε, εισηγητές και τους σκιάδες. Ο κύριος Άλπα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ, κύριε Μηχανικέ. Ε, ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Κύριε Μηχανικέ. Τέτοιε μέρε το μετανιώνει κανεί που δεν έχει πάει πολυτεχνείο και έχει κάνει άλλε σπουδέ στη ζωή του ε, πολύ λιγότερο χρήσιμε. Ε, επανειλημμένα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα και φαίνεται προφανές ότι όλοι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν ένα φυσικό δίλημα που ε, είναι από την ίδια της, ε, τη φύση της καύσης. Θα περιορίσουμε το διοξίδιο του άνθρακα, τα, καυσαέρια ε, και θα χάσουμε σε απόδοση ή το αντίθετο. Ποια είναι η καλύτερη τεχνική λύση για να λυθεί αυτό το δίλημα, γιατί από ό,τι φαίνεται οι δύο αυτοί στόχοι είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Χωρίς μικρόφωνο. Κατά την άποψή μου, ο καλύτερος τρόπος να ε, συγκεραστούν αυτά τα δύο που είναι αντιφατικά έχει γίνει στα βαρέα οχήματα, στα φορτηγά πριν από λίγα χρόνια, που λειτουργούν πάρα πολύ αποτελεσματικά γιατί έχουν υψηλή θερμοκρασία καύσης μεν, ο κινητήρα δηλαδή παράγει πάρα πολλά οξύδια του αζότου, αλλά στη συνέχεια μετά τον κινητήρα ε, έχουν ένα έλεγχο ή ένα είδο ECR ε, στον, ε, στην εξάτμιση και σε αντίθεση με πολλά γεωταχή, γιατί εγώ δεν ξέρω σε καμία περίπτωση τέτοιο. Ε, στα γιοταχή αυτό που σε ενδιαφέρει είναι ένα μικρό το τεπόσιντο της βενζίνης ας πούμε. Τα φορτηγά έχουν σχεδιαστεί για να έχουν σταθερή ταχύτητα και να κυκλοφορούν συνήθως στον ε, αυτοκινητόδρομο. Ενώ στα γιοταχή είναι διαφορετική η κατάσταση. Μπορεί κάποιο να είναι πιο συντηρητικό ή πιο σπορτίφ στην οδήγηση και εκεί μένονται οι ταχύτητες. Ενώ στα φορτηγά είναι πιο εύκολο γιατί σχεδιάζονται για να κινούνται μια συγκεκριμένη ταχύτητα πολύ ε, ώρα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με αυτό τώρα, θα μπορούσατε να μας πείτε κατά την άποψή σας πώς αξιολογείτε το μέλλον της ε, βιομηχανίας της πετρελαιοκίνησης, τον δίζελ δηλαδή θα πρέπει να αντιγράψουμε αυτό που κάνουν τα φορτηγά ή με τη σημερινή τεχνολογία στα ΙΟΤΑΧΗ έχουμε φτάσει στα όρια μας, στα όρια της τεχνολογίας. Ή μπορούμε να φιλοδοξούμε στο μέλλον να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην κατανάλωση καυσίμου και λιγότερες εκπομπές καυσαερίων. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ήταν ενδεχομένω κατά την άποψή σας και με ποιο τρόπο. Όταν λέω ότι μπορεί να λειτουργεί καλά ένα φορτηγό, πρέπει να σκεφτούμε ότι λειτουργεί καλά, όχι όμως τέλεια και η οικονομία που κρύβεται από πίσω είναι κάπως διαφορετική. Υπάρχουν κάποια τεχνικά μέτρα που επιτρέπουν ανακύκλωση των καυσαερίων αλλά και καθαρισμό τους ε, υπό ένα ευρύ φάσμα συνθήκων, αλλά όλα αυτά στοιχίζουν. το πιο ακριβό και πιθανότατα ε, το καλύτερο μέτρο είναι να υπάρχει εξωτερική ανακύκλωση. Δηλαδή να γίνεται αναρρόφηση των καυσαερίων πάλι ε, στον κινητήρα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό. Το πρόβλημα με τους ε, διζελοκινητήρες είναι ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά, αλλά έτσι θα γίνουν πολύ πιο ακριβές, θα γίνουν πολύ πιο ακριβή αυτοί οι κινητήρες, κάτι που θα αποτελέσει πρόβλημα για τα μικρά αυτοκίνητα, τα ΙΟΤΑΧΗ. Μπορεί λοιπόν ε, βαθμιά να αποσυρθούν οι διζελοκινητήρες για τα γιοταχή, για μεγάλα αυτοκίνητα και ε, για τα φορτηγά. Ε, νομίζω ότι οι διζελοκινητήρες είναι η καλύτερη επιλογή. Ευχαριστώ κύριο Σκερπράντη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την εισαγωγή σας και τις πρώτες απαντήσεις που μας δώσατε. Στην προηγούμενη ακρόαση είχαμε εκπρόσωπο από το Ολλανδικό Ινστιτούτο TNO, ο οποίος αρνείται ότι υπάρχει αντιστάθμισμα ανάμεσα στην ε, αποδοτικότητα του κινητήρα και ε, τις εκπομπές οξυδίων του αζότου. Επίσης ισχυρίστηκε ότι δεν είναι απαραίτητο να ανασταλεί η λειτουργία ε, των μηχανισμών ναι, η να μην υπάρξει ζημιά στον κινητήρα. Στην ερώτηση 3 λέτε ότι μετά από ε, ε, εξετάσεις κινητήρων ε, με κάποια κεραμικά τμήματα μπορεί να υπάρξει ε, αύξηση της θερμοκρασίας και να καταστραφεί ο κινητήρας. Ε, αυτό, καταρχάς τι εννοείται με αυτό και πόσο συχνά γίνεται αυτό, μία φορά το χρόνο ή κάθε πέντε λεπτά, διότι αυτό ε, η απάντηση θα δώσει κάπως διαφορετική απόχρωση στο θέμα αυτό. Τα κεραμικά υλικά για ε, τις εξατμίσεις οδηγεί σε αντίσταση σε θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών Κελσίου. Η εξάτμιση ενός διζελοκινητήρα συνήθως ε, δεν ε, φτάνει τέτοιες θερμοκρασίες. Γι' αυτό λέω σε ακραίες περιπτώσεις. Συνήθως η εξάτμιση ε, ενός διζελοκινητήρα φτάνει θερμοκρασίες κάποιων εκατοντάδων βαθμών Κελσίου, όχι όμως χιλιάδων. Σε ε, κινητήρες ε, αερίου, αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί. Επιπλέον θα πρέπει να σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα μεγάλο μέρος του τμήματος επεξεργασίας ε, των καυσαερίων βρίσκεται κάτω από το αυτοκίνητο. Αυτό όμως μπορεί να είναι πιο δύσκολο να γίνει στο μέλλον, διότι ο καταλήτης ACR τοποθετείται πιο κοντά στον κινητήρα. Εδώ υπάρχουν κάποια ε, πλεονεκτήματα, διότι ε, έτσι βρίσκεται πιο κοντά στον ε, κινητήρα, αλλά μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. ο κύριος Κερπράντη, δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει στους διζελοκινητήρες, υψηλές θερμοκρασίες δηλαδή. Επίσης αναφέρεται ότι πιστεύετε ότι μερικές φορές είναι λογικό το, το φάσμα θερμοκρασιών του EGR αλλά λέτε ότι η 70 βαθμοί Κελσίου δεν είναι ρεαλιστική τιμή. Εσείς ε, πού βρίσκετε ότι θα είναι ε, το λογικό φάσμα. Εάν ε, κάνει κρύο, τότε έχουμε πολύ πιο γρήγορη συμπίκνωση των υδρατμών. Οι ε, εμπειρογνώμονες λοιπόν ε, παίρνουν το αυτοκίνητο, πηγαίνουν ε, σε κάποιο δρόμο και κάνουν τις δοκιμές εκεί. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον τα αυτοκίνητα που έχουν πολύ μεγαλύτερο φάσμα θερμοκρασιών και να τα χρησιμοποιήσουμε ως βέλτιστες πρακτικές. Για παράδειγμα, εάν έχουμε παράκαμψη του ψύκτη, μπορούμε να φτάσουμε στις βέλτιστες αυτή τη στιγμή τιμές δηλαδή κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου. Αυτό βραχυπρόθεσμα είναι, πιθανό να, είναι δυνατό να γίνει. πιο μακροπρόθεσμα μπορούμε να πέσουμε και κάτω από το 0. Δηλαδή πιστεύετε ότι το φάσμα 22 με 30 βαθμούς Κελσίου δεν έχει νόημα και πιστεύετε ότι μπορούμε να επιδιώξουμε θερμοκρασίες κάτω των 10 βαθμών, αλλά πιστεύετε ότι με την παρούσα τεχνολογία είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα συγκεκριμένο φάσμα τιμών ε, θερμοκρασίας. Ε, πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε προβλήματα με τις υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες αλλά βέβαια με διαφορετικό σχεδιασμό του συστήματος ε, SCR και έχοντας ένα λογικό φάσμα θερμοκρασιών με παράκαμψη του ψύκτη μπορεί να χαμηλώσουμε τις ε, θερμοκρασίες. Ο κύριος Κερπλάντη, από τεχνικής άποψης, ε, δεν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο αυτό που κάνουν κάποιοι κατασκευαστές αυτοκινήτων να Σβήνει δηλαδή η τεχνολογία για τον ε, καθαρισμό των εκπομπών όταν πέφτουμε κάτω από 20 βαθμούς. Όχι, κατά τη γνώμη μου πολύ νωρίς ε, ε, κλείνει το σύστημα, αναστέλλεται η λειτουργία του. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια, κάποιος τεχνικός λόγος για κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κάρινς, ευχαριστώ πολύ. Πολύ πιο ενδιαφέρον το απόγευμα από ότι φανταστικά διαβάζοντας τις γραπτές σας απαντήσεις. Θα δείτε και από τις δικές μου ερωτήσεις πόσο απέχω από τα τεχνικά και τα τεχνολογικά. Κοιτάω την απάντησή σας στην πρώτη ερώτηση ε, από πλευράς μηχανικής. Μιλάτε για 20.000 ε, πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη και 11 μεγάλες κατηγορίες. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένας κατασκευαστής υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές και υιοθετεί το σύστημα EGR που προτείνεται και το βάζει και στα ΙΟΤΑΧΗ. Από πλευράς τώρα δοκιμών, δεδομένου ότι υπάρχουν τόσα διαφορετικά στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, την ισχύ και ένα σωρό άλλα που δεν θέλουμε να χάσουμε ισχύ από τον κινητήρα, από τελεσματικότητα, αλλά να συγκρατήσουμε την θερμοκρασία, να μην ανέβει πολύ ψηλά, να μην πέσει πολύ μέσα στον κινητήρα, όλα αυτά. Από πλευράς λοιπόν δοκιμών, πώς τα βλέπετε για να εξασφαλίσετε ότι ο κατασκευαστής θα συμμορφωθεί προς τα όσα πρέπει να συμμορφωθεί. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι πάρα πολύ περίπλοκο ε, από πλευράς ε, μηχανικής το ίδιο το λογισμικό. Δεν, όλα αυτά λύνονται με κάποιους πηχαίους τίτλους. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δοκιμή αξιόπιστη. Ε, γιατί υπάρχει μια γενής περιπλοκότητα. Πώς δουλεύουν οι μηχανικοί. Έχουμε ένα στόχο. Και θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Μέσα σε ένα κύκλο. Και αυτό έκαναν αν χρειάζεται μια ρεαλιστική δοκιμή, χρειάζεται να μελετήσουμε όλα τα ενδεχόμενα και όλες τις δυνατότητες. Γι' αυτό θα πρέπει να μελετήσουμε όλες τις καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Και δεν μπορούμε να περιορίσουμε τις μετρήσεις στο, στον ε, κύκλο, ας πούμε. Μισό λεπτό χρειάζεται συνήθως ε, στη θεωρία ε, για να πας από τα 0 στα 50 χιλιόμετρα. Μα κανείς δεν οδηγεί έτσι, δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι ανεδαφικές οι συνθήκες που εκτιμούμε για τον κύκλο μελέτης της δοκιμής που να απέχουν από την πραγματικότητα. Το RD είναι το καλύτερο τεστ, η καλύτερη δοκιμή, δηλαδή ε, real drive Στι συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Δηλαδή αυτό μπορεί να γίνει μάλιστα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενθαρρυντικό αυτό που μας λέτε. Ε, να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση για να βεβαιωθώ ότι σας κατάλαβα καλά. Το ε, Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας μίλησε και για το μέγεθος των κινητήρων και είπε ότι οι μικροί κινητήρες έχουν ε, μεγαλύτερα προβλήματα και στο μέλλον οι μικροί κινητήρες πρέπει να δεχτούν όλη αυτή τη τεχνολογία. Υπάρχουν περιορισμοί και λόγω της φυσικής και μόνο. Ναι, το πρόβλημα της φυσικής δεν είναι βασικό. Το βασικό είναι το πρόβλημα του κόστους. Είναι το οικονομικό. Γιατί είναι υψηλέ οι δαπάνε για να γίνει ο κινητήρα αυτό σε σχέση με το μέγεθό του. Και ε, στη αφορτηγά, α πούμε, στι μεγάλους κινητήρες ή ακόμα για να το τραβήξω παραπάνω σε ένα κινητήρα πλοίου, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτό. Άρα οι καταναλωτέ θέλουν να αγοράσουν και ένα αυτοκίνητο που να είναι φτηνό, αλλά εμείς στην νομοθεσία μας ε, δίνουμε φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα για μικρούς κινητήρες. Αυτό θα είναι τώρα ενθάρρυνση για τις εταιρείε να φτιάχνουν τέτοιους κινητήρες που να μην είναι καλύτερη δυνατή λύση μπορεί να γίνει αυτό, αλλά από την άλλη υπάρχουν τώρα υβριδικοί κινητήρες και προχωράει η τεχνολογία και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με τις αγορές που αναδύονται και με τους μικρούς ε, κινητήρες diesel. Αυτή τη στιγμή είναι πιο ακριβή, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να αυτηνίνουν. Ωραία, ευχαριστώ. Ο κύριος Αρτούκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Δόκτωρ Μπόργκεστ. Ε, χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ και είστε και από την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Αν σας κατάλαβα καλά, γιατί και εγώ δεν είμαι μηχανικός, υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αυτό το παράθυρο, η θηρίδα για τις θερμοκρασίες και κατά την άποψή σας χρειάζεται αυτή ε, η συσκευή ε, ο αναστολής ή διακοπής λειτουργίας και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και είπατε ε, ότι η καλύτερη λύση θα ήταν μια εξωτερική επιστροφή του καυσαερίου, αλλά αυτά θα ήταν πολύ ακριβή. Αν ήσασταν εσεί τώρα νομοθέτης, τι θα κάνατε τελικά, τι θα επιλέγατε ω την καλύτερη λύση και τι θα προτείνατε για να αποτρέψουμε και τις καταχρήσει και να προστατεύουμε και τον κινητήρα. Αν ήμουν νομοθέτης, δεν θα προέβλεπα κανένα ειδικό τεχνολογικό μέτρο, απλώς ε, υψηλά μεν όρια, αλλά στα πλαίσια του εφικτού και ρεαλιστικές δοκιμές. Αυτά, αν κατάλαβα σωστά την ερώτησή σας. Και αυτό φυσικά ε, θα οδηγούσε σε λύσεις από εκεί και πέρα καλύτερες από αυτές που ισχύουν σήμερα κάθε κατασκευαστής θα επιλέξει τον πιο φθηνό δρόμο. Και υπάρχουν δρόμοι πολύ φτηνοί ε, να ξεφύγεις από τις δοκιμές χωρίς να είναι πραγματικά καθαρό το αυτοκίνητο. Για την ομοθετησία λοιπόν χρειάζονται ρεαλιστικές τιμές οριακές και ρεαλιστικές δοκιμές που θα αναγκάσουν τους κατασκευαστές να επιδείξουν δημιουργικότητα και φαντασία και να φέρουν την τεχνολογία αυτή μέσα στα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν απαντώ ακριβώς την ερώτησή σας. Um, Μάλιστα, αυτό που μας περιγράψατε στα γερμανικά ε, το λέμε... Ε, ε, ε, μια, μια μέθοδο για να δικαιολογηθεί αυτή η θηρίδα των θεμοκρασιών και εάν μπορεί να αποφευθεί πώς αποφεύγεται. Αποφεύγεται. Αυτό δηλαδή να γεμίζει κάπνα ο, η εξάτμιση. Αν ελέγχουμε τη θερμοκρασία, δηλαδή να μην πέσει πολύ, αποφεύγεται αυτό σε ένα λογικό πλαίσιο θερμοκρασιών. Γιατί και κάποια στιγμή μείον 20 υπάρχουν θερμοκρασίες ε, που είναι ψυχρές συνθήκες η κίνηση και ο κινητήρας και δεν μπορεί αυτό να αποφευθεί. Κολλάει κάπνα δηλαδή, καπνιά στο κινητήρα και αυτή δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα που υπάρχει. Άρα ε, πρέπει κανείς να συνεχίσει να εργάζεται εκεί και να κάνει έρευνα, ιδιαίτερα η μηχανική. Και έχω και άλλη ερώτηση. Ο Ντόρμπριντ, υπουργό μεταφορών της Γερμανίας, έκανε πρόταση την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο, θα το παρακολουθήσατε, όπου οι ε, συσκευές αυτές αναστολής θα ε, ε, μπορούν να ε, νομιμοποιηθούν γιατί λόγω των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων αυτές είναι αναπόφευκτες. Και ε, πώς το ορίζει αυτό, πώς ορίζεται η πιο πρόσφατη τεχνολογική εξέλιξη. Νομίζω ότι είναι αρκετά ελαστική αυτή η διάταξη, υπερβολικά ελαστική. Δηλαδή δεν συμφωνείτε με κάτι τέτοιο. Ναι, όντω δεν συμφωνώ. Και έχω άλλη μια ερώτηση. Βλέπω ότι είναι προβληματικό ότι και οι δύο πλευρές, και οι κατασκευαστές ε, και οι καταναλωτές, θέλουν ε, να περάσει η δική τους θέση. Δεν ε, θα ήταν χρήσιμο στα υπάρχοντα αυτοκίνητα εφόσον το σύστημα το χειρίζεται ένα λογισμικό Το λογισμικό επίσης να συμπεριλαμβάνεται στην έγκριση τύπου και μάλιστα να παρουσιάζεται το λογισμικό κατά την έγκριση. Η συμπερίληψη του λογισμικού στην έγκριση τύπου είναι προβληματικό θέμα, διότι είναι πάρα πολύ δαπανηρό να αναλύσει κανείς το λογισμικό. Μάλλον δεν θα είναι δυνατόν να αναλυθεί πλήρως, πόσο μάλλον που υπάρχουν διάφορες εκδοχές του λογισμικού για κάθε μοντέλο. Δεν θα είναι εφικτό λοιπόν κάτι τέτοιο. Χρήσιμο όμως θα ήταν δείγματοληπτικά να αναλυθούν κάποιες εκδοχές ε, του λογισμικού και μάλιστα να αναλυθούν πλήρως. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται το λογισμικό που υποβάλλεται να είναι πράγματι το λογισμικό που τοποθετείται στα αυτοκίνητα, διότι αλλιώς μπορεί κανείς να στείλει άλλο λογισμικό για εξέταση και άλλο να βάλει στο αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σχένκε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω διάφορες ερωτήσεις, τις οποίες μπορείτε να απαντήσετε πολύ σύντομα. Είπατε ότι το φάσμα θερμοκρασιών που χρησιμοποιείται από κάποιους παραγωγούς, 20 με 30 βαθμούς Κελσίου, είναι ε, υπερβολικά στενό Μπορείτε να ποσοτικοποιήσετε το φάσμα αυτό και μπορούμε να το ρυθμίσουμε επίσης. Να πούμε δηλαδή ότι από την τάδε μέχρι την θερμοκρασία να μην μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του, του, ε, της συσκευή. Πιο χρήσιμο θα ήταν να γίνουν κάποιες μετρήσεις αναφοράς με όλα τα τεχνικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να εξεταστεί ε, σε ποιες θερμοκρασίες παρουσιάζονται τα προβλήματα. και έτσι θα μπορούσαμε να θέσουμε τις οριακές τιμές σε πολύ ε, στεναρή βάση. Ε, θα μπορούσαμε λοιπόν ε, να θεσπίσουμε ένα φάσμα το οποίο να μην μπορούν να τηρήσουν κάποιοι κατασκευαστές. Ε, ε, μπορούμε να πούμε στους κατασκευαστές ότι μέσα στο φάσμα 0 έως 35 βαθμούς να μην μπορεί να αναστελεί η λειτουργία. να το πω κάπως διαφορετικά. γίνονται δοκιμές και από τους κατασκευαστές, αλλά για να ποσοτικοποιήσουμε το συγκεκριμένο φάσμα θα πρέπει η αξιολόγηση αυτή να γίνει από ε, κάποιον ανεξάρτητο φορέα. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ε, τι φάσμα μπορούμε να πετύχουμε χωρίς ε, ιδιαίτερη προσπάθεια, ενώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις νέες τεχνολογίες. Εάν λοιπόν ε, εξετάσουμε τι είναι δυνατόν, τότε θα έχουμε χρήσιμα στοιχεία, αλλά αυτά θα πρέπει να καθοριστούν από κάποιον ανεξάρτητο φορέα. Ο κύριος ε, Χένκελ, μιλήσαμε πολύ για αυτά τα φάσματα θερμοκρασιών. Υπάρχει κάποιο άλλο φάσμα, για παράδειγμα το υψόμετρο ή η υγρασία. Ναι, το υψόμετρο είναι κάτι το οποίο πρόσφατα συζητήθηκε πολύ. διότι υπάρχει ο μηχανισμός που αραιώνει τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ε, όταν ε, όμως οδηγούμε σε υψηλό υψόμετρο ε, είναι ήδη πιο αραιή η ατμόσφαιρα και έτσι εάν αραιώσουμε περαιτέρω τον αέρα αυτόν τότε θα έχουμε εθάλη και έτσι μπορούμε να έχουμε ένα φάσμα ατμοσφαιρικής πίεσης όπου να μην υπάρχει πρόβλημα, αλλά και πάλι θα πρέπει να προσέξουμε πού θα θέσουμε τα όρια. Μπορούμε να θέσουμε τέτοιο φάσμα ώστε ακόμα και ψηλά στις Άλπεις ε, να, μπορεί να, ε, να μπορούμε να οδηγούμε χωρίς ε, πολλά καψαέρια. Ή άνω των 700 ε, ε, μέτρων ε, να υπάρχει ανασταλή του μηχανισμού. Χρειάζεται δηλαδή να θεσπίσουμε και ένα φάσμα για το υψόμετρο, για την υγρασία τι ισχύει. Για την υγρασία δεν βλέπω να υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Ο κύριος Χένκελ, επόμενη ερώτηση. Η FEV, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ε, διαπίστωσε ότι η ποιότητα του αέρα επίσης ε, επηρεάζει τα αποτελέσματα των ε, ελέγχων, του, του καυσίμου. Ε, σίγουρα η ποιότητα του καυσίμου επηρεάζει την, τις εκπομπές. Δεν ε, μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τι θα μπορούσε να κάνει ο νομοθέτης, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το σκεφτούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευχαριστώ πολύ. Είπατε τα πράγματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε με τον τρόπο αυτό που θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε. Η πρώτη μου ερώτηση έχει σχέση με αυτά που είπατε τον Φεβρουάριο του 2016. Είχατε πει ότι δεν εμπιστεύετε τόσο πολύ τους κατασκευαστές. Αυτό λοιπόν που ονομάζουμε Dieselgate ή σκάνδαλο της Volkswagen ε, αποκάλυψε κάτι το καινούριο για σας ή υποπτεύεστε και τώρα και τότε ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται δεν είναι οι καλές, οι σωστές. Για δέκα χρόνια έλεγα στους φοιτητές μου ότι μια μεγάλη ανοησία γίνεται και ότι οι κύκλοι δοκιμών στην ουσία γίνονται με συνθήκες ιδιαίτερα βελτιωμένες. Ικανοποιήθηκα λοιπόν όχι από το Dieselgate αλλά για το ότι δημοσι... μου έκανε εντύπωση βέβαια το ότι δημοσιοποιήθηκε αυτό το 2015 και όχι νωρίτερα. Ε, ευχαριστώ για την απάντηση. Κάποιοι άλλοι κατασκευαστές, όχι η Volkswagen υποχρεωτικά, ήρθαν, ε, σας πλησίασαν για να εξηγήσουν αυτά τα οποία κάνουν και μπόρεσαν να σας δώσουν ε, με πληροφορίες τις οποίες πιστεύετε ότι είναι έγκυρες. Όχι, δεν μου έδωσαν πληροφορίες. Έδωσαν κάποιες εξηγήσει. Been... σε σχέση με το SDS, αλλά οι πληροφορίες αυτές ήταν πολύ γενικού τύπου. Δεν εξήγησαν πραγματικά το το οποίο συμβαίνει. Τελευταία ερώτηση. Είναι δυνατόν για τους κατασκευαστές να αλλάζουν τις ρυθμίσεις των υπολογιστών των αυτοκινήτων έτσι ώστε τα συστήματα EGR ή ρύθμισης καυσαερίων να σταματούν τη λειτουργία τους. Ή μόνο οι κατασκευαστές των υπολογιστών μπορούν να το κάνουν αυτό. Απαιτείται ένα ειδικό λογισμικό, ε, θεωρείται ότι το λογισμικό αυτό λειτουργεί παραπλανητικά, απαιτείται για να υπάρξει παρέμβαση μια απλή ρύθμιση ή ο κωδικός πηγής του υπολογιστή. Εγώ είπα δύο διαφορετικούς τρόπους για να ξεπερνιέται αυτή η δυσκολία. Ο παραδοσιακός τρόπος είναι ότι ο προμηθευτής ή boss σαν παράδειγμα δίδει ε, ε, το λογισμικό χωρίς τα δεδομένα. Τα δεδομένα τα βάζει ο κατασκευαστής, τα όρια τα βάζει ο κατασκευαστής και μετά μένει πάντα ανοιχτό το σύστημα εκτός και αν ξεπεράσει κάποια όρια. Οι κατασκευαστές βέβαια είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τα όρια όπου αυτοί νομίζουν πιο σωστό, όπου τους βολεύει καλύτερα. Το δεύτερο μοντέλο είναι ο παραγωγός να δώσει μία μονάδα ηλεκτρονική, ένα ETU, με ένα ουδέτερο software, στην ουσία μια, ένα, ένα σύστημα λειτουργίας Linux, και ε, με νέες μορφές αρχιτεκτονικής μπορεί ο κατασκευαστής να αναπτύξει από μόνος του τους κωδικούς του, τους κωδικούς πηγής και να χρησιμοποιήσει και εργολάβους έτσι ώστε να μπορέσει το σύστημα αυτό να δουλεύει. Η κυρία Κονέτσνα. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά για τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που έχετε και την πραγματογνωμοσύνη και την τεχνογνωσία, του εξή. Μας είπατε ότι εσείς θα θέλετε υψηλές οριακές τιμές και ρεαλιστικές αλλά και ρεαλιστικές δοκιμές. Σωστά ε, το λέω. Ε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σήμερα στην Ευρώπη αυτά είναι ανεδαφικά. Δηλαδή έχουμε βάλει προδιαγραφές και οριακές τιμές ανέφικτες με βάση τη σημερινή τεχνολογική δυνατότητα. Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, μακροπρόθεσμα θα μπορούσα να φανταστώ να τεθούν αυτά τα όρια ακόμα πιο χαμηλά, αλλά οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ρεαλιστικές, αλλά στην πράξη κανένας ε, δεν ενδιαφέρεται για αυτές. Προτεραιότητα λοιπόν για μένα είναι να εφαρμόσουμε τις τιμές που ισχύουν αυτή τη στιγμή και αργότερα να κάνουμε το επόμενο βήμα να προχωρήσουμε σε πιο χαμηλές τιμές. Όπως σας έγραψα όμως, μου φαίνεται σημαντικό πρώτα να εφαρμόσουμε τις τιμές αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο εργαστήριο, αλλά και στο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Θα... Ήθελα επίσης να ρωτήσω κάτι που απαντήσατε στις γραπτές ε, ή και στις προφορικές σας απαντήσεις. Ε, λέτε ότι οι κατασκευαστές ε, δεν είναι αρκετά καινοτόμοι. Είπατε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις νέες ιδέες. Γιατί πιστεύετε ότι δεν αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες που μπορούν και στα πιο μικρά οχήματα να οδηγήσουν σε μείωση των εκπομπών με, χαμηλότερο, με χαμηλότερη τιμή. Στο παρελθόν δεν υπήρχε η ανάγκη για τους κατασκευαστές να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικές ε, τεχνολογίες, διότι μια χαρά πέρασαν από τους έλεγχους μέχρι τώρα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όσον αφορά τον κανονισμό για τις Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς ε, τις ώστε να, έχει, να συμμορφώνεται με όλες τις τιμές ε, και με τα σωματίδια και με τα άλλα αέρια. Ε, καταφέραν λοιπόν να πετύχουν τη σωστή ισορροπία ε, στο εργαστήριο, αλλά γνωρίζουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουν τις ε, ακριβείς τιμές ε, για τις ε, πραγματικές συνθήκες. Αλλά ο κύκλος δοκιμών, ο κύκλος οδήγησης δεν απαιτεί κάτι τέτοιο και γι' αυτό δεν έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη καλύτερων συστημάτων. Στις γραπτές σας απαντήσεις λέτε το εξής, ότι οι αρχές ελέγχου χρειάζονται περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο δεν θα πρέπει να συνδέεται άμεσα ή έμεσα με ε, λόμπι. Πώς το βλέπετε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα ελέγχων. Εγώ μηχανικός είμαι. Γι' αυτό, για το θέμα αυτό, θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Προσωπικά πιστεύω πως ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρίντα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, μιλήσαμε για ε, το φάσμα των ε, θερμοκρασιών. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, θερμοκρασία κίνησης του κινητήρα. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες θερμού κινητήρα στις εκπομπές σε σχέση με ψυχρό κινητήρα. Ε, με ψυχρή κίνηση θα πρέπει να είναι πιο χαμηλές ή πιο ε, ψηλές ε, οι τιμές. Γενικά, απαιτούνται υψηλότερε θερμοκρασίε, δηλαδή ο θερμό κινητήρα θα πετυχαίνει καλύτερε τιμέ. Και η επόμενη μου ερώτηση είναι Ε, ότι στη Γερμανία διαπιστώθηκε ότι σε 48 από 53 αυτοκίνητα διαπιστώθηκε ακριβώς το, το αντίθετο ότι με ψυχρή εκκίνηση ήταν πιο χαμηλές οι τιμές. Ε, αυτό πώς μπορείτε να το εξηγήσετε. Από τεχνικής άποψης ε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Κάτι πάει στραβά εδώ. Επίσης, ε, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ε, αναφέρει στην έκθεσή της για το Όπελ Zafira ότι ε, πληρεί την τιμή για την ψυχρή κίνηση, κατά την θερμία κίνηση, οριακά καλύπτει τις τιμές. Αν κατάλαβα, δηλαδή θα έπρεπε να είναι χαμηλότερες οι τιμές κατά την εκκίνηση με θερμοκινητήρα. Εκτός μικροφώνου. Εάν ε, δεν παρεμβαίνει το λογισμικό, τότε θα έπρεπε να μειώνονται οι τιμές και όχι να αυξάνονται. Το συμπέρασμα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας ήταν ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω έλεγχοι, ε, αρκεί απλά η Όπελ να κάνει τις σχετικές ρυθμίσεις δεν συμφωνείτε με ένα τέτοιο συμπέρασμα. Μικρόφωνο χρειαζόμαστε για τη μετάφραση. Είπατε λοιπόν στις γραπτές σας απαντήσεις ότι η χαμηλότερη αποτελεσματικότητα του συστήματος AGR κατά τις χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να εξηγηθεί με λιγότερες εκπομπές μικροσωματιδίων. αλλά αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει στην περίπτωση των αυτοκινήτων που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν. Κάθε αυτοκίνητο θα πρέπει να ε, πληρεί τις ε, τιμές για τα μικροσωματίδια. Ωστόσο, ε, το φίλτρο δεν μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα κατά 100%. μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα. 50% θα πρέπει να ε, γίνει διάκριση ανάλογα και με το μέγεθος ε, των ε, μικροσωματιδίων. Διότι μπορεί να περνούν τα πολύ μικρά σωματίδια παρόλα αυτά, δηλαδή παρά το φίλτρο, μπορεί να υπάρχει ανάγκη να έχουμε μικρό, λιγότερη εκπομπή από τον κινητήρα ή να έχουμε φίλτρο ώστε να έχουμε αποτελεσματικότητα 100%. Κάτι ακόμα. Είπατε ότι δεν υπάρχει τεχνολογική αιτιολόγηση ε, για την ε, αναστολή του συστήματος SCR ε, κατά ταχύτητες άνω των 145 χιλιόμετρων την ώρα. Υπάρχει θεωρητικά κάποια εξήγηση και είναι ρεαλιστικό Ε, να μην ζητάμε καν Δυστυχώ Δυστυχώς ε, δεν ξέρω τι γνωρίζει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, θα ήθελα πάρα πολύ όμω να το ξέρω. Ειλικρινά δεν μπορώ να σα δώσω απάντηση. Ε, καλά, αυτό το πρόβλημα καταρχήν δεν θα πρέπει να είναι διαφορετικό. Ο κατασκευαστή να λέει σε τι χρησιμεύει αυτό το σύστημα που αναστέλει τη λειτουργία και μετά να εγκριθεί. Ναι, αν ήμουν εγώ ομοσπονδιακή υπηρεσία θα ήθελα να γνωρίζω γιατί φτιάχνουν τέτοιες συσκευέ έχουν δώσει μια εξήγηση και μια αιτιολόγηση που δεν είναι πάντα ε, κατανοητή. Ε, το ECR ε, βάζει ένα κατόφλι ταχύτητας, εγώ θα το έκανα διαφορετικά, αντίστροφα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Γιατί έγινε αυτό, αλλά δεν τους γνωρίζω. Και μπορεί να είναι αποχρόντες και θεμητοί, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ θα μετρούσα τη θερμοκρασία και ενδεχομένως και την ταχύτητα ε, αλλά όχι ως αποκλειστικό κριτήριο. Ευχαριστώ. Η κυρία Εύη. Ε, Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ενδιαφέρουσα, χρήσιμη αλλά και περίπλοκη τεχνικά. Μία ερώτηση λοιπόν για τα τεστ αυτά, τα RDE, όπως έγιναν πρόσφατα δεκτές ε, το 2001, το προσωρινό και το 5 το τελικό. Μπορείτε να με βεβαιώσετε ότι αυτοί οι παράγοντες συμβατότητας ή συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα γενναιόδοροι και τελικά μη απαραίτητοι υπό το φως των τεχνολογιών που μας παρουσιάσατε λίγο πριν. Λέτε για τις ισχύουσες διατάξεις σήμερα. Για τις πρακτικές μάλλον που χρησιμοποιούνται σήμερα και το νέο RDE με τους νέους αυτούς παράγοντες ε, ε, συμμόρφωσης 2,1 και 2,5. Πιστεύετε ότι είναι ιδιαίτερα γενναιόδοροι οι παράγοντες αυτοί. I think we cannot build cleaner cars Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να χτίσουμε αυτοκίνητα καθαρά. Απαιτείται μια μεταβατική φάση με υψηλότερες σταδιακά αξίες αλλά θα πρέπει η μεταβατική περίοδος να είναι η συντομότερη δυνατή. Ε, Μια άλλη ερώτηση. σχετικά με τον κύκλο δοκιμών Άρτεμις. αν είχαμε σήμερα ήδη σε λειτουργία αυτά τα τεστ για την έγκριση τύπου και όχι το ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών, αν το είχαμε αυτό, πιστεύετε ότι θα είχαμε σε κυκλοφορία σήμερα αυτοκίνητα τα οποία θα εξέπεμπαν λιγότερο, πιο καθαρά αυτοκίνητα δηλαδή. η έλλειψη δημιουργικότητας τελικά είναι συνέπεια εν πολλής από τον παρόντα κύκλο δοκιμών που δεν απαιτεί να γίνονται ιδιαίτερες προσπάθειες. Με το νέο κύκλο τώρα έχουμε το New LTC και έχουμε επίσης και τις, ε, το RDC. Οι διαφορές ανάμεσα στους δύο αυτούς κύκλους είναι ότι περιλαμβάνει ευρύτερα ε, πιο δυναμικά παραδείγματα οδήγησης, τύπους οδήγησης. Ενώ στο παρελθόν εμέναμε σε περιβάλλοντα εργαστηρίου. Νομίζω λοιπόν ότι ο συνδυασμός των δύο νέων αυτών τύπου κύκλων μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε καθαρότερα αυτοκίνητα. Μία τελευταία ερώτηση για την δυνατότητα ανείχνευσης των μηχανισμών παραπλάνησης που να εναλλάσσουν σε εργαστηριακό περιβάλλον από τον ένα κύκλο στον άλλο αλλάζοντας ταχύτητες και χρόνο οδήγησης. Πιστεύετε ότι αυτό θα διευκολύνει να ανοιχνεύονται τα συστήματα παραπλάνησης. Εγώ μίλησα για την έλλειψη δημιουργικότητας. Ίσως όμως μερικές φορές να φτάνουμε σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδα. Υπάρχει δημιουργικότητα στην εφαρμογή κάποιων μηχανισμών παραπλάνησης πολύ ευφυών που δεν είναι δυνατόν να ανοιχνευθούν εύκολα με τους διάφορους κύκλους. Υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι μηχανισμοί πάρα πολύ απλοί. Όταν ας πούμε είναι αναμένη μηχανή με τον ίδιο μέσον όρο θα έλεγα κύκλου δοκιμών αλλά αντί να γίνεται σε ένα, σε ένα test bench, σε μια επιφάνεια δοκιμών, να γίνεται στην οδήγηση, σε πραγματικές συνθήκες. Ίσως όμως να υπάρχουν και άλλα τέτοια συστήματα τα οποία να είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοιχνευθούν. Κύριε καθηγητά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Ε, αισθάνομαι λίγο σαν να ξανακάθισα στα φοιτητικά έδρανα. Κατάλαβα μερικά πράγματα. Νομίζω όλοι μας μας βοήθησαν ε, να καταλάβουμε περισσότερα σήμερα. Όταν μιλούσατε για αυτή τη θηρίδα των θερμοκρασιών που χρειάζεται για την πίεση και γιατί χρειάζεται να μπορεί να διακόπτεται η λειτουργία ε, ενός συστήματος λόγω ατμοσφαιρικής πίεσης και τα λοιπά. Πρόσφατα για το Opel έγραφε ένα άρθρο, ε, ε, ένα μεγάλο γερμανικό περιοδικό, χωρίς να δίνει την ίδια εξήγηση που δώσατε εσείς τώρα. Εσείς ως επιστήμονας αυτή τη στιγμή πώς αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Γίνονται διάφορες ε, συμβουλές και οδηγίες και δεν περιμένουν κάποιοι να απαντήσει η Opel. Γιατί και εγώ μηχανικός είμαι και ε, αισθάνομαι ότι ε, σπέβδουμε να καταδικάσουμε κάποιους πριν να απαντήσουν, πριν έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν. Φυσικά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαντούν οι ενδιαφερόμενοι. Ε, γιατί εδώ σε μια περίπτωση που είχαμε συζητήσει, που ήταν το όριο Ταχύτητα για το ECR μπορεί να υπάρχει λόγος και θα ήθελα να το μάθω. Ας του αφήσουμε ναι, την ευκαιρία να απαντήσουν, να δώσουν τους λόγους που του οθούν να κάνουν κάποια πράγματα και βλέποντα και κάνοντας. Ευχαριστώ για την απάντηση. Έχω και δεύτερη ερώτηση. Σπούδασα λίγα χρόνια και μετά εργάστηκα περισσότερα στην αγορά και υπάρχει εξή διαφορά. Ε, ως μηχανικός ε, στο Πανεπιστήμιο θεωρούσα ότι μπορούσαμε να βρούμε λύση για τα πάντα. Είμαστε ευφυείς, είμαστε ξύπνοι, είμαστε δημιουργικοί και φάνταστοι και θα τα λύσουμε όλα. Αλλά πολύ συχνά δεν ψάχναμε πόσο κοστίζει η λύση. Ε, στην αγορά κοιτάνε και λίγο πόσο κάνει αυτό, γιατί όταν παράγεις και κατασκευάζεις αυτοκίνητα, κοιτάς και τι... Ε, είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης, πόσο βαθιά να βάλει το χέρι στη τσέπη. Είπατε ότι υπάρχουν δυνατότητε, αλλά πολλά από αυτά είναι δαπανηρά. Ε, αναφερθήκατε και σε μια θερμοκρασία τάξη των μείων 20 βαθμών ε, Κελσίου, αλλά τώρα ξέρουμε ότι είναι διαφορετική η τάξη μεγέθους. Όχι σε ευρώ, σε ποσοστά μπορείτε να μας πείτε πάνω κάτω μια τάξη μεγέθους που κινούμαστε. Ένα σύστημα ελέγχου των καυσαερίων, ε, πόσο θα κρύβαινε το αυτοκίνητο, κατά πόσο θα αυξανόταν η τιμή εάν χρησιμοποιούσαμε την τεχνολογία που θα μας χρειαζόταν και την οποία συζητάμε όλη τόση ώρα η τέλεια λύση είναι πάρα πολύ ακριβή για την εσωτερική συγκράτηση των καυσαερίων. Είναι με, με διάφορες βαλβίδες και τα λοιπά και τελικό κόστος θα ήταν κάποιες εκατοντάδες ευρώ για τον ε, ε, κατασκευαστή και σε μικρό αυτοκίνητο, σε μικρό κινητήριο θα ήταν σημαντικό το κόστος και για τον πελάτη. Αλλά μπορούν να υπάρχουν ε, ε ή εγκαταστάσεις ε, ψήξης πιο φτηνές, που δεν είναι ιδεώδεις. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση Δηλαδή πόση δουλειά χρειάζεται άνα κινητήρα, άνα ε, αυτοκίνητο για να εγκατασταθεί και μετά το κόστος της έρευνας και της ανάπτυξης που μπορεί να είναι φάπαξ, ε, αλλά υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικά ε, αυτοκίνητα. Ευχαριστώ. Κύριε Σπεντιτσίνη. Ευχαριστώ. Οι εξηγήσει σας ήταν σαφείς, συγκεκριμένες. Ε, ας πούμε ότι για 72 ώρες έχετε την δυνατότητα εσείς για να πάρετε μέτρα για την καταπολέμηση των νόξ. Το πρώτο θέμα στο οποίο θα παρέμβετε είναι η κύκλη δοκιμών που δεν είναι ρεαλιστική. Κατάλαβα σωστά. Ο κατασκευαστής χρειάζεται κάποιο χρόνο για να προσαρμόσει την τεχνολογία σε αυτόν τον πιο σοβαρό κύκλο δοκιμών. Αυτός όμως είναι καλός τρόπος να επιβάλλουμε ρεαλιστικές τιμές. Δεν είμαι βέβαιος αν αυτό απαντάει στην ερώτησή σας. Μάικρο, μάικρο, μάικρο. Ε, Εν μέρη, πιο ρεαλιστική κύκλη δοκιμών και αυτό θα μειώσει και το κόστος. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητάμε εδώ και εβδομάδες, έχουμε πάρα πολλά επίπεδα δυνατότητας παρέμβασης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε. Λοιπόν, ποιοι είναι οι κύκλοι που πρέπει να ακολουθήσουμε αν θέλουμε εμείς να ελέγξουμε αυτά τα επίπεδα πιθανής παρέμβασης. Domanda uh, semplice. semplice. Uh, I would attend. Δεν είναι ναι. πολύ εύκολο. Ναι. Δεν είναι πολύ... Δεν είναι πολύ εύκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ανέφερα διάφορα τεχνικά μέτρα. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών μέτρων ε, στη διάθεσή μας για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Μερικά μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα, ενώ άλλα απαιτούν πολλές έρευνες ακόμα. Και αυτό είναι ο λόγος που λέω ότι εάν ελαχιστοποιήσουμε τα παραθυράκια Εάν επιβάλλουμε δηλαδή τις τιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ασκούμε πίεση στους κατασκευαστές ώστε να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό είναι παρόμοιο με αυτό που αναφέρατε κι εσείς. Πολλά είναι δυνατόν να γίνουν. Δεν ε, υπήρχαν όμως οικονομικά κίνητρα για τους κατασκευαστές να κάνουν ε, πράγματι το δυνατό. Sì. Il punto di partenza sono sempre i cicli Πάντα πάντως στο σημείο εκκίνησης παραμένουν, παραμένουν οι κύκλοι δοκιμών. Έχουμε όμως ανάγκη από πραγματικούς, ρεαλιστικούς κύκλους δοκιμών, γιατί αλλιώς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα τη απουσία δεδομένων. Αποτέλεσμα. Η κυρία Τούν ε, Χόνστάιν. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή και ε, για μένα είναι πολύ χρήσιμο σήμερα που έμαθα ότι το Ασάφενπουργκ βρίσκεται στη Βαβαρία. Αλλάζει κάπως την εικόνα που είχα για τη Γερμανία αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για τα αυτοκίνητα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα κατασκευάσουμε με τρόπο πιο καθαρό από τη μία μέρα στην άλλη. Τα μικρά διζελοκίνητα οχήματα μπορεί βαθμιά να αποσυρθούν από την αγορά. τι πιστεύετε ότι θα αντικαταστήσει τις σημερινές τεχνολογίες. Ποια τεχνολογία θα αντικαταστήσει τα μικρά διζελοκίνητα οχήματα. Ποια είναι η τεχνολογία που είναι πιο πιθανό να επιβληθεί στην αγορά. θα γίνουν πιο, ακριβές οι μικρές, θα γίνουν πιο οι μικροί διζελοκίνητοι κινητήρες στο μέλλον. Απ' την άλλη θα γίνουν πιο οικονομικοί οι υβριδικοί κινητήρε. Αυτή τη στιγμή ο διζελοκινητήρα είναι πιο οικονομικό από τον υβριδικό, αλλά θα αυξηθεί η τιμή για του διζελοκινητήρε εάν ε, εισάγουμε επιπλέον μέτρα. Ενώ υπάρχει η πτωτική τάση για τους υβριδικούς κινητήρες και τελικά ο ίδιος ο κατασκευαστής αυτοκινήτων θα αποφασίσει Ωραία, φτάσαμε τώρα ε, στο μηδενικό σημείο. Δεν χρειάζεται η νομοθεσία να κάνει τίποτα. Ο κατασκευαστής θα επιλέξει την ε, καλύτερη λύση για να πετύχει τις ε, απαιτήσει στην καλύτερη τιμή. Ο υβριδικός κινητήρας λοιπόν είναι η μία πιθανότητα. Επίσης, ε, στο παρελθόν ε, το πλεονέκτημα του διζελοκινητήρα σε σχέση με τον κινητήρα ε, με τους άλλους κινητήρες ε, ήταν η αποδοτικότητα, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από άλλους παράγοντες. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε τελικά κινητήρες βενζίνης. Από την άλλη, όσο πιο αποδοτικοί γίνονται οι κινητήρες βενζίνης, ε, τόσο πιο πολύ αρχίζει και μοιάζει ε, ο τρόπος ε, καύσης με τον διζελοκινητήρα. Το μέλλον λοιπόν θα δείξει πώς θα χειριστούν οι κατασκευαστές ε, τις ε, τεχνολογίες αυτές. άλλε εναλλακτικές λύσεις είναι άλλα καύσιμα. Για παράδειγμα, στην ε, Σκανδιναβία χρησιμοποιούν αέριο σε κάποιε περιπτώσει. και κατά την καύση αερίου. Δεν λύνει κανεί το πρόβλημα οξυδίων του αζότου, έχει όμω κανεί λιγότερα μικροσωματίδια. Και έτσι μπορεί κανεί ε, να προσαρμόσει ε, τον κινητήρα ώστε να μειωθούν και οι εκπομπέ ε, οξυδίων του αζότου. Ε, ευχαριστώ κύριε Βονταλόν. Ευχαριστώ. Στην αρχική σας τοποθέτηση μας παρουσιάσετε τις διάφορες δυνατότητες τεχνολογικές για να βελτιωθεί το κάθε διαφορετικό σύστημα, κάθε συσκευή. Βέβαια μας είπατε ότι το κάθε σύστημα έχει το κόστος του. Και μας θυμήσατε ταυτόχρονα τις Ηνωμένε Πολιτείες, τα αυτοκίνητα ε, που πολλούνται εκεί είχαν ε, ε, το σύστημα ECR για να ανταποκρίνονται στις αυστηρές προδιαγραφές των Ηνωμένων Πολιτείων. Πέρα από το κόστος αυτά τα συστήματα, οι συσκευές από πλευράς, μεγέθους και βάρους μπορούν να μπουν και σε μικρά αυτοκίνητα δίζελ ε, ή από πόσα κυβικά και πάνω. Δεν είναι μόνο το κόστος, είναι και το μέγεθος του κινητήρα. Ε, ακούστηκε από πολλούς ότι είναι περίπλοκο σε ένα μικρό αυτοκίνητο να μπουν όλες αυτές οι συσκευές ε, που Ε, δεν επιτρέπουν την ακύρωση και το, το λογισμικό το απατηλό. Από τεχνική σκοπιά είναι ακόμα πιο εύκολο να γίνει καθαρό ένα μικρό αυτοκίνητο από ότι ένα μεγάλο SUV. Ε, είναι οικονομικό περισσότερο το πρόβλημα για τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Γιατί όταν είναι μικρό το αυτοκίνητο και μικρός ο κινητήρας, ε, ποσοστία είναι μεγάλο το κόστος. Αν για παράδειγμα παίρνεις ένα αυτοκίνητο 8.000 ευρώ ή μάλλον 80.000 ευρώ, δεν σε νοιάζει αν αυξηθεί η τιμή κατά 1.000 ή 2.000 ευρώ. Αν αγοράσει ένα αυτοκίνητο 15.000 ευρώ μπορεί για κάποιον και τα 1.000 και τα 2.000 να είναι δαπάνη. Άλλο που ρωτήσατε, πώς έχει η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, για την Αμερικανική αγορά, πολλοί κατασκευαστές έχουν πιο προηγμένα συστήματα καυσαερίων, ε, δηλαδή καθαρισμού από τα καυσαέρια, αλλά και πιο ακριβά. Ας πούμε, μία εταιρεία, ε, δεν χρειάζεται να πω το όνομα για να μην κάνω διαφήμιση, αλλά μια εταιρεία έχει αγοράσει ένα πολύ καθαρό σύστημα πολύ καθαρό. Ε, έχει φέρει στην αγορά την αμερικανική καθαρούς διζελοκινητήρες, ε, ακριβούς όμως αρκετά. Και από την άλλη μπορούμε να δούμε ότι ορισμένοι κατασκευαστές έχουν μεγάλα προβλήματα να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ΗΠΑ Υπάρχει και άλλος Γερμανός κατασκευαστής που προσπαθεί να διεισδύσει στην Αμερικανική αγορά και δεν θα πρέπει να λεσμονούμε και το λεγόμενο Dieselgate, ότι αποκαλύφθηκε ή ανακαλύφθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χένκελ. Ε, όλοι έχουμε ενθουσιαστεί ε, από τη νέα λύση πλέον, ε, το ε, δε, που μας προτείνεται, αλλά έχει και ένα μειονέκτημα. Κάποια στιγμή γερνάνε και τα αυτοκίνητα diesel. Ε, τώρα αν δοκιμάζεται ε, το νέο σύστημα Real Drive σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, τι γίνεται μετά από 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια. Θα κυκλοφορεί το αυτοκίνητο ακόμα καθαρό αυτό είναι πολύ σωστό που ρωτάτε. Με το νέο σύστημα αυτό των δοκιμών δεν μπορεί να διαπιστωθεί αυτό και υπάρχουν και προβλήματα. Σας είπα για τα καυσαέρια ε, ε, υπάρχει ένας σένσορας και ε, αυτός ο αισθητήρα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου γιατί μπορεί να στρέφει τα αέρια σε λάθος κατεύθυνση. Οι κατασκευαστές ε, παίρνουν ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας. Τώρα, κατά πόσο ο καταλήτης αυτός θα παραμείνει καθαρός καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του αυτοκινήτου, θα πρέπει να γίνονται συνεχώς δοκιμές. Μπορεί να γίνει αυτό στο εργαστήριο, αλλά είναι τεχνητές οι συνθήκες αυτές και όχι πραγματικές. Θα μπορούσε να γίνει όπως γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε να αποσύρονται αυτοκίνητα από την κυκλοφορία και να ελέγχονται μετά. Άρα θα πρέπει να, γίνει και αυτό σε ένα τέτοιο σύστημα ως δοκιμή. Μάλιστα και άλλη ερώτηση. Τώρα μιλήσαμε για defeat ε, devices, συσκευές ε, ε, εξαπάτησης και η Mitsubishi πλέον και η Suzuki πιάστηκαν στα πράσα, όχι με λογισμικά αλλά και με το υλικό. αποκαλύφθηκε αυτό, βγάλανε κάποια πιο ελαφριά αυτοκίνητα στην αγορά, αποκαλύφθηκε αυτό στην Ιαπωνία και παρετήθηκε μετά από λίγες μέρες ο πρόεδρος της εταιρείας, σε αντίθεση με τη Γερμανία. Τα, ε, ξέρετε εσείς αυτά είναι γνωστά τα προβλήματα για σας. Ναι. Στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι αυτό πιο πολύ και όχι στα νόξ, ότι κάποια στιγμή πρέπει να εγκριθεί ο τύπος σύμφωνα με τη μάζα του αυτοκινήτου και την αντίσταση στον αέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολοι υπολογισμοί, πάρα πολύ περίπλοκοι ε, που ανοίγουν μεγάλο περιθώριο σε σφάλμα και μπορεί να είναι και ε, επίτηδες αυτό εσκεμμένο. Παράδειγμα, για τα ελαστικά τα φουσκώνουν περισσότερο. Κάνουν ε, ε, διάφορα κόλπα και τεχνάσματα στο εργαστήριο, κολλάνε ε, διάφορες σχισμές του, του ελαστικού μία ταινία για να κάνουν τις μετρήσεις, αλλά δεν μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο έτσι ένα αυτοκίνητο με τα λάστιχα πειραγμένα. Να ρωτήσω διαφορετικά. Ο κύριος Ντάνιελ Λάγκε και ο Φίλιξ Τουίν έχουν δώσει διάφορες εξηγήσεις σε εφημερίδες και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας έχουν δώσει πολλές πληροφορίες και μάλιστα ο κύριος Λάγκε είναι προσκεκλημένος μας σήμερα τους ε, τελευταίους μήνες διαπίστωσα ότι αυτοί οι δύο κύριοι ήταν ε, οι πρώτοι και μάλλον οι μόνοι που μπόρεσαν ε, να διαπιστώσουν τροποποίηση του λογισμικού. Είχαν κάποιες υποδείξεις παράνομης συμπεριφοράς. Πολλά χρόνια εργάζονται στον τομέα αυτών. Εσείς όταν μιλάτε με τους φοιτητές σας, ή με άλλους ε, λάβατε πληροφορίες με τέτοιες πρακτικές, σχετικά με τέτοιες πρακτικές. Στον κλάδο αυτόν είναι πολύ γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι ο κύκλος δοκιμών δεν είναι ρεαλιστικός και ότι ο καθένας βελτιστοποιεί ε, τα αποτελέσματα για το αυτοκίνητό του και δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στο δρόμο. Αυτό εδώ και πολύ καιρό γίνεται στον κλάδο αυτόν και το γνωρίζει ο, ο καθένας που εργάζεται ε, σε αυτόν τον τομέα. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συσκευές αναστολής, αυτό είναι νέα πληροφορία. Σας ευχαριστώ για την απάντηση αυτή. Το πρώτο μέρος της απάντησής σας είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες και οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται σε αυτές. Από τη μία δηλαδή έχουμε τις συσκευές αναστολή, αλλά από την άλλη προσαρμόζεται κανείς στο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν είναι ε, παράνομο. Μόνο οι συσκευές ε, αναστολή ε, είναι παράνομες. Ε, ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς ε, παράνομο, αλλά ο, ο καθένας ε, δίνει την ερμηνεία που θέλει στους κανόνες. Ε, και εγώ αν ήμουν κατασκευαστής, μάλλον το ίδιο θα έκανα. Μέχρι... Ε, μάλλον εάν ο νομοθέτης μου λέει ότι μη σε νοιάζουν αυτές οι τιμές, τότε ουσιαστικά ε, με ενσαρρύνει να κάνω το αντίθετο και ακριβώς ε, λόγω του ε, ε, πολύ ασαφούς ορισμού του συστήματος αναστολής παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Ερτούκ, κύριε Μπόργκεστ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και για μη ειδικού. Τώρα, ξαναδιάβασα αυτή τη διαφάνεια που μας δείξατε, αυτό το σχεδιάγραμμα και αν κατάλαβα καλά αυτό τώρα που σας δείχνω τι είναι. Είναι ο έτσι, από εδώ φεύγουν τα καυσαέρια και επαναχρησιμοποιούνται. Δηλαδή τη θερμοκρασία τη χρησιμοποιούν, τη θερμότητα για θέρμανση. Και ε, μερικά φεύγουν από, το, από την εξάτμιση από τον καταλήτη. Ναι, 35, ένα τμήμα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ωραία. Ε, ερωτώ τώρα. Τι διακόπτεται το LNTCR ανάλογα με τα συστήματα. Ε, προστατεύεται ο κινητήρας όταν διακόπτει τη λειτουργία ενός συστήματος μετά τον κινητήρα πίσω, τον, πίσω από τον κινητήρα στην εξάτμιση. Τι προστασία κινητήρα είναι αυτή. Έχει νόημα για τον κινητήρα αυτό. Για τον κινητήρα τον ίδιο αυτό που συμβαίνει από πίσω του δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι τι, πώς ορίζεται ο κινητήρας. <laughs> κινητήρας δηλαδή είναι μόνο εκεί που καίγεται το καύσιμο ή το σύνολο. Ε, ε, κινητήρε εσωτερικής καύσης και τα καυσαέρια. Για τον κινητήρα αυτό καθ' αυτό τον πυρήνα του είναι μάλλον αδιάφορο και τελείω άσχετο το τι συμβαίνει μόλι φύγουν από εκεί τα καυσαέρια. Ο κ. Γκερμπράντι. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας είπατε ότι οι κατασκευαστές δεν ενδιαφέρονται για να φτιάξουν καθαρότερα αυτοκίνητα αλλά ενδιαφέρονται για να ξεγελάσουν τους κύκλους δοκιμών. Και οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σαν στόχο ακριβώς αυτό, το να ξεγελάσουν τον κύκλο δοκιμών. Σωστά κατάλαβα? Ακριβώς λέει ο μιλητής. Αυτό υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία τελικά που έχουν οι κύκλοι. Είπατε επίσης ότι δεν εκπλήσεστε για όλα αυτά, Εκπλήσεστε όμως γιατί ήρθαν στην επικαιρότητα και φανερώθηκαν μόνο το 15. Εσείς γνωρίζετε την κατάσταση. Θεωρείτε ότι οι δημόσιες αρχές ήταν ενήμερες για το τι συμβαίνει. Όχι μόνο για τους μηχανισμούς παραπλάνησης, αλλά για το ότι οι επιχειρήσεις, οι αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν σαν στόχο το να ξεγελάσουν τον κύκλο δοκιμών. Οι Αμερικανικές αρχές τα ήξεραν αυτά. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες είτε δεν ήξεραν ή λένε ότι δεν ήξεραν. Προσπάθησαν να μην ξέρουν μάλλον. Ας πάρουμε μια περίπτωση μελέτης στη Γερμανία εσείς σαν καθηγητής είσαστε σε επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα συζητάτε τα θέματα αυτά. Είχατε τη δυνατότητα να το συζητήσετε αυτό τα τελευταία χρόνια με εκπροσώπους του δημοσίου τομέα. Όχι. Διαβάσατε οτιδήποτε προέρχεται από δημόσια πηγή, από δημόσια αρχή η οποία να αποδεικνύει ε, σε εσά ότι τα γνώριζαν αυτά. Μπορούσε να διαβάσει κανείς για δοκιμές από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από ιδιωτικές οργανώσεις, στις οποίες οι δημόσιες αρχές δεν αντέδρασαν. Εσείς πιστεύετε ότι για λόγους επιβολής και προστασίας ενός κοινού αγαθού όπως ε, η καθαρότητα του αέρα θα έπρεπε να παρέμβουν ε, οι δημόσιες αρχές. Επαναλαμβάνω, υπήρχε μια κάποια γενική αντίληψη γύρω από όλα αυτά ότι υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στους κύκλους δοκιμών και τις πραγματικές εκπομπές. Πιστεύετε ότι οι αρχές θα έπρεπε να παρέμβουν νωρίτερα. Ναι νομίζω. Ο κύριος Ζάλμπα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μία ερώτηση σε επίπεδο τεχνικό. Η μεταβατική περίοδος για να πετύχουμε τους νέους στόχους των εκπομπών Euro 5, Euro 6 είναι επαρκής και τι γίνεται στις άλλες αγορές όπως η ΙΠΑ και η Απονία. αν και έχω εργαστεί με τους Ιάπωνες, δεν ξέρω πώς δουλεύει η Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή. Στις Ηνωμένε Πολιτείες δεν έχουν υπάρξει μεγάλες περίοδοι μεταβατικές. Αν όλα πάνε καλά, οι κύκλοι αυτοί δεν θα έπρεπε να είναι καν απαραίτητοι. Αλλά ζητήθηκαν, εν για να πετύχουμε τις απαιτήσει. Στις Ηνωμένε Πολιτείες πάντως οι κατασκευαστές γνωρίζουν τι θα συμβεί εάν προσπαθήσουν να εξαπατήσουν. Και με λίγες εξαιρέσεις έχουν πετύχει τα όρια. στις Ηνωμένε Πολιτείες λοιπόν δεν έχουν υπάρξει μεταβατικές περίοδοι. Ευχαριστώ. Μια άλλη ερώτηση. Μου φαίνεται ότι είστε υπέρ των υβριδικών. Τα υβριδικά λειτουργούν με κινητήρες βενζίνης ε, εσωτερικής καύσης. Θα ήταν δυνατόν με την παρούσα τεχνολογία να υπάρξει υβριδικό και με πετρελαιοκινητήρες. Είναι δυνατόν να υπάρξουν υβριδικά με ε, δίζελ, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχεις και το αυξημένο κόστος του πετρελαίου και το αυξημένο κόστος του υβριδικού ηλεκτροκινητήρα. There are Υπάρχουν κάποια Λοιπόν, υπάρχουν κάποια υβριδικά με πετρέλαιο, αλλά είναι εξαίρεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως αυτό θα μπορούσε να γίνεται και γίνεται και ίσως να είναι σωστό. Νομίζω πάντως ότι δεν είναι μια, μεγάλη, μια λύση με μεγάλη εμβέλεια εφαρμογής. Η κυρία Σεντέρ. Eh, Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί είχα άλλη ανηλυμένη υποχρέωση ε, και δεν άκουσα την παρατήρησή σας, την τοποθέτηση μάλλον και θέλω να σας ρωτήσω το εξή επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ε, τον κλάδο που μας απασχολεί, τι πιστεύετε, πώς να το διατυπώσω τώρα. Τα μέτρα που εμείς απαιτήσαμε από τον κλάδο Πού οδήγησαν επιταχύθηκαν οι κύκλοι εφαρμογών των μέσων σε τέτοιο σημείο και βαθμό που αυτό να προκάλεσε κάποια δημιουργική και φάνταστη λύση εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί το είπατε κι εσείς, για κάποια προϊόντα υπάρχουν κύκλοι παραγωγής και δοκιμών που πρέπει κανείς να προβλέπει σε βάθος χρόνου τις εξελίξεις και μάλιστα για διάφορες κατηγορίες σε μια χώρα ας πούμε έχουμε μικρά και μεσαία γιοταχή, όχι τα μεγάλα, στα αφήσουμε τα μεγάλα. Ένα από τα ε, μέτρα που προτείνεται είναι πιο φτηνό, μάλλον πιο ακριβό από τα άλλα. Άρα ακριβένει και η τελική τιμή για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα αν καταστεί υποχρεωτικό αυτό το σύστημα στη μεταβατική περίοδο μέχρι να βρούμε το ιδανικό αυτοκίνητο που ούτε ρηπαίνει, ούτε καυσαέρα βγάζει, ούτε μυρίζει, ούτε τίποτα. Πόσο θα πήγαινε. Θα μπορούσε να φθηνίνει η παραγωγή αν είναι μαζική, αν υπάρχει οικονομία κλίμακας. Αυτό το AdBlue για πιο μικρά και μεσαία αυτοκίνητα είναι δυνατό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε πετρελαιοκίνητα οχήματα. Και μια άλλη ερώτηση. Ακούγεται η πρόταση τώρα να μεταβούμε ε, σε πιο μικρά αυτοκίνητα, μέχρι τρία λίτρα κατανάλωσης. Γίνεται αυτό κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να συμφωνήσουμε έτσι ώστε τα μέτρα και η δοκιμή να είναι πραγματική και όχι εικονική, όχι στο εργαστήριο, ακόμα και αν ρηπαίνουν. Αντί να ψάχνουμε διάφορες φόρμουλες για να ξαναφανίσουμε τη ρήπανση. Γίνεται λόγος για τα βεζινοκίνητα τώρα να πάμε σε κινητήρες κάτω των τριών λίτρων. Τι προτείνετε. Μα ο καθηγητής τώρα έχει δέκα δεύτερα να απαντήσει θεωρητικά, αλλά θα του δώσω λίγο παραπάνω χρόνο. ναι, It's It's okay. Yes, Κύριε καθηγητά μου. Come to your first question. Όσον αφορά την πρώτη σας ερώτηση, είναι δυνατόν αυτές οι νέες επιπλέον τεχνικές λύσεις ε, στο μέλλον να είναι λιγότερο δαπανηρές. Κάποιες, ναι, αναφερθήκατε στο SCR. Ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω πως όχι, διότι ο καταλήτης είναι πολύ ακριβώς ε, και υπάρχει ένα σύστημα αν, αντλίας ε, και δοσολογίας. δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος. Ίσως όμως να αναπτυχθεί μια τελείω νέα αρχή για τους καταλήτε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως άλλες τεχνολογίες τι οποίες ανέφερα. που απαιτούν κάποια προσπάθεια για την ανάπτυξή τους. Για παράδειγμα, ανέφερα ότι μπορεί να έχουμε νέα υλικά τα οποία ε, να αποτρέπουν ε, το, το βούλωμα του κινητήρα. Και κάτι τέτοιο θα μπορούσε ενδεχομένω ε, να παραχθεί με οικονομικό τρόπο. Και άλλο παράδειγμα. Υπάρχει ένας κατασκευαστής ε, που έχει αυτοκίνητο στην αγορά με διπλή εξάτμιση. Ε, ανακύκλωσης ε, και μπορεί κανείς να έχει εξωτερική ανακύκλωση των καυσαερίων. Μπορεί κανείς έτσι να μπορέσει να μειώσει τις εκπομπές. Αυτό συνδέεται με τα οξύδια του αζότου. Εάν διαπιστώσουμε ότι ε, αυτό το σύστημα ε, SCR χαμηλής πίεσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ε, με τρόπο που να χαμηλώνονται οι εκπομπές μπορεί στο μέλλον να το αντικαταστήσουμε ε, να αντικαταστήσουμε το σύστημα υψηλής πίεσης με σύστημα χαμηλής πίεσης σε ανάλογη τιμή όμως και να γίνουν έρευνες στο τομέα αυτό. Χρειάζεται δηλαδή μία φορά να επενδύσουμε στο θέμα αυτό και να δούμε αν λειτουργεί. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κιλιώνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω, κύριε Πόρκεστ. Εγώ μεγάλωσα κοντά σε ένα γκαράζ και θα ήθελα να γνωρίζω εάν μπορούμε να έχουμε εκ των υστέρων προσαρμογή των αυτοκινήτων, διότι έχουμε... Ε, μεγάλο στόλο αυτοκινήτων που χρειάζεται εξοπλισμό μείωσης των εκπομπών. Θα ήταν ε, μάλλον πιο έξυπνο να διορθώσουμε τα αυτοκίνητα που υπάρχουν ε, αντί να περιμένουμε όλος ο κόσμος να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο. Πώς βλέπετε λοιπόν ε, την δυνατότητα με μετεξοπλισμού των αυτοκινήτων. διότι νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει αναφερθεί ως λύση μόνο για φορτηγά και λεωφορεία. Αλλά αναπτύσσονται τεχνολογίες ε, μείωσης της ρήπανσης. Πώς θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι ότι λέμε συνέχεια ότι η έρευνα απαιτεί χρόνο, η τεχνολογία είναι δαπανήρη. Εάν θεσπίσουμε αυστηρά όρια, εάν έχουμε απαιτητικό κύκλο δοκιμών, τι μεταβατική περίοδο χρειάζεται η βιομηχανία για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσει. Νομίζω ότι είναι σημαντικές οι δύο που θέσατε. Καταρχάς όσον αφορά τον μεταξοπλισμό. Ανάλογα με τη χώρα, ε, έχουν ε, τα αυτοκίνητα κύκλο ζωή 10 χρόνια. Έχουμε άλλες ε, μηχανές γεωργικές, οικοδομικές με πολύ μακρύτερη ζωή, 20, 30, ίσως και 50 χρόνια. Ο μετεξοπλισμός λοιπόν θα ήταν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Από τεχνικής άποψης είναι όμως δύσκολο να γίνει διότι θα πρέπει να διεισδύσει κανείς ε, στη μηχανή, στον έλεγχο του κινητήρα. Θα πρέπει δηλαδή να αντικαταστήσει κανείς όλο το σύστημα ελέγχου του κινητήρα, κάτι που είναι δύσκολο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αδύνατο, αλλά είναι δύσκολο να γίνει. Θα σας παρακαλούσα να, να επαναλάβετε τη δεύτερη ερώτησή σας. Πολύ σύντομα, λέει η Πρόεδρος. Ναι, θα είμαι σύντομη. Τι χρόνο πιστεύετε ότι θα χρειαστεί η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις για να προσαρμοστούν εάν θεσπίσουμε νέα πολύ αυστηρά όρια και έχουμε καλό και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων στο μέλλον. Εάν δηλαδή οι πολιτικοί λάβουν τις σχετικές αποφάσεις. Τη δεκαετία του 70 συζητήθηκε να ε, εισαχθούν καταλήτες ε, τριπλή για τους διζελοκινητήρες. Ε, τότε υπόθηκε ότι ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Θεσπίστηκε όμως ο νόμος και ξαφνικά λειτουργούσαν, βρέθηκαν καταλήτες που να λειτουργούν. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να πει κανείς πόσο χρόνο θα απαιτήσει κάτι τέτοιο και πόσο θα στοιχήσει. Νομίζω ότι αν υπάρξει πίεση είτε από την πλευρά της αγοράς είτε από την πλευρά της νομοθεσίας, πολύ συχνά είναι δυνατόν να εφαρμόσει κανείς νέα τεχνολογία μέσα σε τρία χρόνια. Αλλά βέβαια αυτό εξαρτάται από την πολυπλοκότητα εδογίας. Ευχαριστώ πολύ. Ρέντα παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα, δώστε το παράδειγμα. Κύριε ε, Δόκτωρ Μπόργκε, στις γραπτές σας απαντήσεις αναφέρετε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η δημοσιοποίηση ε, του λογισμικού να είναι σκόπιμη και να βελτιώσει ε, την εφαρμογή του νόμου. Το ένα είναι η τεκμηρίωση του software, του λογισμικού. Μια τέτοια τεκμηρίωση αυτόματα θα περιείχε τέτοιες πληροφορίες ε, για ποιο σκοπό έχει δημιουργηθεί αυτό το λογισμικό και θα πληρούσε την προϋπόθεση ότι ε, κάθε ε, μηχανισμός αναστολής λειτουργίας μιας άλλης ρύθμισης θα μπορούσε να εγκριθεί, δηλαδή με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Στην τεκμηρίωση και στα χαρακτηριστικά θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι η σωστή. <laughs> γιατί μπορεί να καταθέτουν κάποια στοιχεία αλλά να μην είναι το λογισμικό αυτό που εγκαθίσταται στο αυτοκίνητο. Να είναι ακριβή και ειλικρινή τα στοιχεία. Είναι πολύ περίπλοκο αυτό. Ακόμα και μικρή αλλαγή στο ε, λογισμικό μέσα σε μια ώρα χρειάζεται κανείς να το ψάξει ε, μία με δύο εβδομάδες για το τι επιπτώσεις θα έχει στο λογισμικό. Και εκεί ε, η τεκμηρίωση βοηθάει πολύ τα documentation, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αλλά να είναι η σωστή. Και ένας κατασκευαστής είχε και μια ακουστική λειτουργία κάποτε υποτίθεται. Αυτή όμως η ακουστική λειτουργία είχε άλλο τελείω σκοπό από το να ε, βελτιώνει το θόρυβο. Και αυτός που διαβάζει την τα στοιχεία, την τεκμηρίωση, θα πρέπει να καταλαβαίνει τι κρύβεται από πίσω και τι θέλει να πει ο ποιητή. Το τύφνο, ε, ε, ε, ο αρμόδιο φορέας στη Γερμανία που κάνει τους ελέγχου στο ΚΤΕΟ, είπε ότι θα θέλαμε να μάθουμε την τεκμηρίωση, αλλά ε, κάπου δείχνουν ένα πείσμα. Οι, οι κατασκευαστές σου λένε έχουμε πνευματικά δικαιώματα και είναι πνευματική μα ιδιοκτησία. Υπάρχουν θέματα εκεί εμπορικού απορρίτου που πρέπει να προστατεύεται κανονικά κάθε ένας ε, που έχει να κάνει με εμπορικό απόρριτο στη βιομηχανία υπογράφει αντίστοιχη συμφωνία και αυτό ελέγχεται και, και επίσης εάν άλλος ε, φορέας, ο Prüfnor, Prüfsüd στη Γερμανία, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι δεν θα έρθει ο επόμενο κατασκευαστή και ε, να πει τι έχουμε εδώ, να το πάρω και εγώ να το βάλω στα αυτοκίνητά μου. Αυτό το πράγμα λύνεται. Αυτό το κάνει και ο προμηθευτής. Κάποιες εταιρείες που δουλεύουν για πολλούς κατασκευαστές και παράγουν εξαρτήματα δεν πάει να ε, μαρτυρήσει το μυστικό του ενός κατασκευαστή στον άλλον. Λύνονται αυτά τα ζητήματα εχημήθειας και απορρίτω. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, καθηγητά που τα εξηγήσατε και τα καταλάβαμε και εγώ που είμαι μια απλή κοινωνιολόγος. Τα κατάλαβα. Οι πολύ επεξηγηματικέ οι απαντήσεις σας, μπορεί να έρθουν και άλλες γραπτές ε, ερωτήσεις και θα σας παρακαλούσαμε να τι απαντήσετε γραπτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και απαντήσατε στι ερωτήσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σα. like our... Θα ήθελα να περάσουμε στην τελευταία για σήμερα κρόαση και ελπίζω να μπορέσουμε να τηρήσουμε και την πειθαρχία και το ωράριο. Um, Παρακαλώ καθίστε. Κύριε Ντάνιελ Λάγκε, είστε διευθύνων σύμβουλος του Faster IT που είναι μια γερμανική συμβουλευτική εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών για το management και τα ηλεκτρονικά. Έχετε 20 χρόνια εμπειρία στην αυτοκινητοβιομηχανία για τη στρατηγική ε, επικοινωνίας και ε, γενικότερα στα ηλεκτρονικά στις τηλεματικές ας πούμε στην εταιρεία BMW και σε άλλες εταιρείες είστε παραπάνω από εμπειρογνώμων για να απαντήσετε στις δικές μας ερωτήσεις έχετε απαντήσει γραπτός και ο κύριος Φέλιξ Ντόμπελ που έχει εργαστεί στην Bosch για τον έλεγχο καυσαερίων συνεργάστηκε μαζί σας για να απαντήσετε τις ε, ερωτήσεις, αλλά αποφασίσαμε στους συντονιστές μετά την ακρόαση αυτή ε, να υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις και στον κύριο Ντόμπερ και προς εσάς. Εντάξει, αν χρειαστεί αυτό και κρυθεί απαραίτητο. Καταρχάς σας καλωσορίζω στη συνεδρίασή μας και σας δίνω αμέσω το λόγο για να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή. Παρακαλώ πολύ. Um, thank you much for the... Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να σας ε, απευθύνω το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και ελπίζω να μπορέσω κατ' λίγο να συνεισφέρω. Είμαι μηχανικός, ε, είμαι όμως ε, ασχολούμαι και με θέματα στρατηγικής μετά από πρακτική. Κάποιοι μηχανικοί ήταν αυτοί οι οποίοι έφεραν στην επικαιρότητα α, την ιστορία του Dieselgate και ήταν οι μόνοι οι οποίοι προσπάθησαν εξ αρχής να διαφωτίσουν το κοινό για το περιεχόμενο της προσπάθειας παραπλάνησης του και τι επίσης έγινε και ίσως ακριβώς μπορώ να βοηθήσω στο να πω πώς θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια απάτη έχουμε να κάνουμε με μία δραστηριότητα οικονομική η οποία η παραγωγή αυξάνεται συνεχώς. Τα αυτοκίνητα γίνονται συνεχώς πιο μεγάλα, πιο πολυτελή και πιο ακριβά. Οι αυτοκίνητοβιομηχανίες είναι σαν δεινόσαυροι οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένους τομείς τους οποίους προσπαθούν να ελέγξουν. Καταλαβαίνετε ότι αν ακολουθούσαμε τη λογική της παραγωγής ε, ενός CPU για ένα υπολογιστή, οι τιμές των αυτοκινήτων θα ήταν πολύ χαμηλότερες σήμερα. Δεν υπάρχει εξήγηση λοιπόν γιατί τα αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο ακριβά. Ακούσαμε στην αρχή της παρουσίασης ότι για να μπορέσει κανείς να επιλέξει το πιο αποδοτικό σύστημα εξατμίσεων κοστίζουν 600-700 ευρώ. Έξω από την είσοδο εδώ θα δείτε ανθρώπους που προσπαθούν να σας εντυπωσιάσουν με τα αυτοκίνητά τους χωρίς οδηγό. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα οικονομική για να ελεγχτούν καλύτερα τα καυσαέρια, κάτι το οποίο ίσως να μην έχει γίνει ακόμα. Τώρα, οι δεινόσαυροι αυτοί έχουν συγκεκριμένες ε, διαδικασίες, δεν αλλάζουν τον κωδικό συμπεριφοράς, τον κώδικα συμπεριφοράς τους σε σχέση με την παραγωγή τους. Οι περίπλεκες ε, διαδικασίες χαρακτηρίζουν επίσης και τις ανταλλαγές εγγράφων και πληροφοριών μεταξύ τους. Ε, κανένας κωδικός δεν θα αλλάξει από την BOS αν δεν υπάρξει ένα αίτημα για την αλλαγή. Υπάρχουν θέματα αν θέλετε ε, συνεπειών νομικών υποχρεώσεων, υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες υπογράφονται από τους διαχειριστές. Οι αλλαγές αυτές ε, ε, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και μέσα σε 4 με 6 εβδομάδες καταλήγουν στην τελική τους μορφή στα διοικητικά συμβούλια. Σε αυτές λοιπόν τις εταιρείες μαμούθ δεν συμβαίνει τίποτα χωρίς να ενημερώνεται η κορυφή τους. Έτσι γίνονται αντικείμενο διαχείρισης. Φυσικά το βασικό κριτήριο είναι το κόστος. Αυτό ακούσαμε και από τους άλλους ομιλητές. Λοιπόν, ή θα υπάρξουν ε, ε, διαδικασίες ε, που ακολουθούνται και οι οποίες χαμηλώνουν το κόστος, ή αλλιώς θα αποτύχουν στην ευθύνη που έχουν να είναι κερδοφόρα η επιχείρηση και να μην βγει κάποιος να πει ότι με κορόιδευσε η επιχείρηση αυτή με ό,τι συνέπειες. Λοιπόν, υπήρχε περίπτωση κάποιοι μηχανικοί να απέκρυβαν την πραγματικότητα σε τεχνικό επίπεδο από την ηγεσία της επιχείρησης. Όχι βέβαια, ένας μηχανικός ηλεκτρολόγος δεν έχει κανένα συμφέρον να κρύβει την κατάσταση από τους ανωτέρους του. Έτσι και αλλιώ ένα πολύ μικρό κομμάτι του μισθού του ανταποκρίνεται στη, ε, στο επίπεδο της μετοχής της επιχείρησης ε, στα χρηματιστήρια. Συνεπώς λοιπόν τα εισοδήματα αυτών έχουν σχέση ακόμα και από τις προβλέψεις τις οποίες ε, η επιχείρηση χρησιμοποιεί για να μπει σε μια συγκεκριμένη αγορά. Έτσι λοιπόν ε, θα έπρεπε οι πολιτικοί όλοι να επιθυμούν και εσείς θα πρέπει να μειώσετε τα κίνητρα για αυτούς τους ανθρώπους τις ηγεσίες των επιχειρήσεων ε, Πρέπει να έχουν κίνητρα λοιπόν και να μην μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι άδικο. Αν σαν παράδειγμα οι αμοιβέ των στελεχών, των ανωτάτων είναι ένας πολλαπλασιαστής των αμοιβών των εργαζομένων ανάλογα με την απόδοση της επιχείρησης, τότε τα πράγματα θα είχαν καλύτερες εξελίξεις. Αν μιλάμε μόνο για την τιμή της μετοχής, τότε στην ουσία η κατάσταση δεν θα αλλάξει και καθηγητές όπως ο προηγούμενος ομιλητής θα σας λένε ότι είναι θέμα κόστους γιατί τα πράγματα δεν αλλάζουν. Λοιπόν, τόσοι άνθρωποι ήξεραν, γιατί δεν έλεγαν τίποτα τόσα χρόνια. Εδώ υπάρχουν δύο απαντήσεις και δυστυχώς και οι δύο δείχνουν προς τις δικές σας κατευθύνσεις. Πρώτον, δεν υπάρχει προστασία για τους whistleblowers, για τους καταδότες δημοσίας ωφέλειας. Ε, κοιτάξτε, ε, αν κάποια πληροφορία θα έσωζε εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους από θανάτους, ασθένειες κτλ. Αλλά θα εγκινδύνευαν τη δουλειά τους και τη ζωή τους. Αν τους προστάτευε η δημόσια προσοχή και ο τύπος, τότε ε, ίσως οι εταιρείε αυτές ε, να είχαν ε, οδηγηθεί και σε πτώχευση. Κοιτάξτε το Snowden. Δεν τολμάμε καν να του χορηγήσουμε άσυλο εμείς σαν Ευρωπαίοι λοιπόν έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε για να ζητήσουμε από άλλους να είναι πιο ειλικρινείς, να έχουν περισσότερο θάρρος. Αν θέλουμε οι άλλοι να έχουν θάρρος, εσείς δώστε το παράδειγμα σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένας άλλος λόγος για τους οποίους οι κανονισμοί αυτοί και οι διαδικασίες παραπλάνησης δεν ανακαλύφθηκαν νωρίτερα ε, αναφέρθηκαν από τον προηγούμενο ομιλητή. Το θέμα είναι ότι αυτός ο νέος ευρωπαϊκός κύκλος δεν είναι νέος, είναι από το 80, αναδιοργανώθηκε το 1997 με τεχνολογία που έχει ξεπεραστεί πάρα πολύ και η βιομηχανία ήξερε ότι δεν ήταν αντιπροσωπευτικός αυτός ο κύκλος. Έπρεπε να βελτιστοποιήσει κανείς το αυτοκίνητο για τη χρήση του οδηγού και για τη χρήση του τεστ. Αν αρχίζουμε να, να παρεμβαίνουμε στο εργαστηριακό περιβάλλον των τεστ, τότε το παιχνίδι αρχίζει να χοντρένει. Νομίζω ότι ο κύριος Χένκελ μας έδωσε ε, και άλλα παραδείγματα ότι είχαν φουσκώσει τα λάστιχα τόσο πολύ που ήταν έτοιμα ε, να σκάσουν, αλλά υπήρχε πολύ μικρή επιφάνεια ελαστικού ε, τριβής πάνω στην άσφαλτο, οπότε όλα πήγαιναν πιο γρήγορα, ε, χρειαζόντουσαν λιγότερη δύναμη για να το κάνουν και η κατανάλωση ήταν πολύ χαμηλότερη. Όλες αυτές οι μικρές προδοσίες είναι πολύ γνωστές. Η ICCT είπε ότι οι μελέτες για τις επιδόσεις των αυτοκινήτων, τα λεγόμενα DIN και είδαν ότι όλοι ε, δίνουν στοιχεία τα οποία δεν είναι απόλυτα αξιόπιστα. Κάποιοι λένε τα πράγματα όπως περίπου είναι και το 15-20% δεν λένε πραγματικά την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία θα κοροϊδέψεις και εσύ με τη σειρά σου τον επόμενο πελάτη όταν πουλήσεις το αυτοκίνητό σου γιατί έτσι και αλλιώς τα στοιχεία που έχουν οι αρχές δεν είναι τα σωστά. Θα πρέπει οι νόμοι να γίνονται σεβαστοί, θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες για οποιονδήποτε τους, παρε... τους παραβαίνει. Είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι ε, είτε ζητώντας μη ρεαλιστική ε, τιμή για κάποια προϊόντα κτλ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω τελειώνοντας είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να μπαίνουμε εμείς σε λεπτομερέστερες κάθε φορά α, λεπτομέρειες. Δεν είναι σωστό να ζητάτε συνέχεια περισσότερες τεχνολογικές λεπτομέρειες. Μην είστε υπερπαρεμβατικοί, μην ζητάτε όλο και περισσότερους και πιο καινούριου τύπους καταλητών. Μην ακολουθείτε αυτόν τον αγώνα στους εξοπλισμούς. Δώστε κατευθυντήριες γραμμές, βάλτε τις κατευθυντήριες γραμμές στην νομοθεσία. Πώς θα πρέπει να είναι οι, ε, μορφές ελέγχου των εκπομπών, τι είναι αποδεκτό σε επίπεδο και αφήστε τους κατασκευαστές να σας δώσουν τις σωστές τεχνικές λύσεις. Μην ρυθμίζετε τις λεπτομέρειες αλλά το τελικό αποτέλεσμα στα πλαίσια φυσικά ενός συστήματος που να ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μια βασική ιδέα εδώ για να είμαστε διαφανείς και αποτελεσματικοί, γιατί να μην ελέγχει κανείς το θέμα αυτό όχι μόνο από πλευράς αρχών, αλλά και από πλευράς πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδιαφερόμενες υποχρεώσεις που θέλουν να κάνουν μετρήσεις και αν ξεπερνάμε τα όρια τα οποία επιτρέπονται, τότε να ζητούμε από τον κατασκευαστή να μας εξηγήσουν. Αν οι εξηγήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τότε θα πρέπει να υπάρξει ένα πολύ σημαντικό πρόσημο. Αν υπάρξει αυτό μία φορά δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ πια. Συμπερασματικό λοιπόν να είναι υπεύθυνο το management των επιχειρήσεων για αυτές τις διαδικασίες. Προστατεύσε τους καταδότες δημοσίας ωφέλειας Ξεφύγετε από την υπερβολική παρέμβαση στις ρυθμίσεις ε, όπως επίσης ε, και ε, να πρέπει να ορίζετε τους στόχους, τους κανονισμούς, αλλά όχι εσείς να προδιαγράφετε τη δουλειά των μηχανικών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι αυτός ο ρόλος σας και έναν τέτοιο αγώνα θα τον χάνετε συνέχεια όποτε τον κάνετε. Θέλουμε σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο αμέσως στους δύο εισηγητές, ο κύριος Κερπράντη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Λάνγε, για την διαφωτιστική παρουσίασή σας. Αδράξατε την ευκαιρία να κάνετε και μία έκκληση για τον Έντουαρτ ε, Snowden μπορεί και να συμφωνώ μαζί σας. Αναφερθήκατε στην ευθύνη της ε, διεύθυνση των επιχειρήσεων. Ζητήσαμε τη συμβουλή σας, επειδή είσαστε ειδικό ε, στην πληροφορική και στο λογισμικό για, για τους κινητήρες. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που αναπτύσσουν το λογισμικό αυτό. Οι προμηθευτές, ε, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, ο προγραμματιστής. Τελικά όμως κάποιος διευθυντής είναι υπεύθυνο. Υποθέτω ότι αυτό είναι ο κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Ναι, πράγματι είναι ο κατασκευαστή του αυτοκινήτου και πάντα υπάρχει ειδικό διευθυντή για το ECU, υπάρχει ένα ε, υπεύθυνο για τον κινητήρα, υπάρχει ένα υπεύθυνο για το μοντέλο που χρησιμοποιεί το κινητήρα. Στην Volkswagen, για παράδειγμα, αυτοί ήταν οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την εταιρεία μετά ήταν αυτοί που είχαν υποχρέωση λογοδοσίας και η Volkswagen ε, προφανώς ε, θεώρησε ότι δεν ε, είναι σε θέση να τους διατηρήσει στις θέσεις τους και να τους υπερασπιστεί. Εσείς νομίζω κάνατε reverse engineering, δηλαδή προσπαθήσατε να ανακατασκευάσετε το λογισμικό. Εξετάσατε τον ε, εξοπλισμό και βρήκατε πολλά πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Εάν δούμε το πώς ε, οι αρχές ε, θα πρέπει να επιβάλλουν τον νόμο, πιστεύετε ότι θα πρέπει να έχουν την εντολή να κάνουν κάτι τέτοιο. Στην εισαγωγή σας είπατε ότι πρέπει να μετακινηθούμε Προ ένα σύστημα συμμόρφωση και επεξήγηση. Ε, ή χρειαζόμαστε και τα δύο. Νομίζω ότι όταν γίνεται η έγκριση τύπου ενός οχήματο, ε, θα πρέπει να ε, λαμβάνουν οι αρχές τα, τα στοιχεία του αυτοκινήτου που είναι σε αυξανόμενο βαθμό λογισμικό. το η δουλειά που έκανε ο Φίλιξ ε, που είχε να κάνει και με την αντιγραφή του λογισμικού ήταν και θέμα τύχης. Πρέπει να είναι κανείς τυχερός ε, για να βρει το σύστημα αναστολής. Ε, βέβαια είναι πιο εύκολο όταν ξέρει κανείς τι κάνει αυτό στη Volkswagen για παράδειγμα. Αλλά αν μας δώσει κανείς το ECU ενός άλλου κατασκευαστή και μας πει βρείτε το σύστημα αναστολής θα κάτσουμε να δουλέψουμε τρει με έξι μήνες και μπορεί να το βρούμε ή όχι. Αλλά το ότι δεν το βρούμε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εγώ λοιπόν θα το έκανα αντίστροφα. Ε, όταν δίδεται η έγκριση τύπου που ο κώδικας ε, που ε, επιτρέπει την ε, λειτουργία του κινητήρα θα πρέπει να υποβάλλεται στους, στις αρμόδιες αρχές ώστε να μπορεί κανείς να αντιγράψει το αυτοκίνητο και το λογισμικό. Και όταν υπάρχουν προβλήματα έχει κανείς ε, τα στοιχεία αυτά και τα εξετάζει είτε δημοσίες είτε αναθέτοντα σε κάποιον συγκεκριμένο. Δεν το κάνει κανεί όμω αυτό αυτομάτω, διότι είναι πολλή δουλειά. Το κάνει κανεί μόνο όταν συμβεί κάτι Για παράδειγμα, δηλαδή, αν παρακολουθεί κανείς ε, την απόδοση ε, του αυτοκινήτου στα χέρια του καταναλωτή, ε, αν όλα λειτουργούν καλά, τότε δεν χρειάζεται να δούμε πόσο το προγραμματίσανε. Εάν όμως όχι, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει κάποια βλάβη, κάποιο λάθος ή υπάρχει εσκεμένα κάποιο σύστημα αναστολής. Ευχαριστώ πολύ Τελευταία μου ερώτηση τότε είναι η εξή. Ε, εσείς ε, όπως ε, και ο καθηγητής Μπόρκε, είπατε ότι πιο πολύ ασχολούνται οι κατασκευαστές αυτοκινήτων με την απάτη κατά τον κύκλο δοκιμών παρά με την απόδοση του αυτοκινήτου στον δρόμο. Συμφωνείτε, εμείς απλά να θέτουμε τα πρότυπα και να εναπόκειται στους κατασκευαστές ε, να τα πληρούν. Έχουμε κάποιους ε, γενικούς... Ε, συμφωνείτε να έχουμε κάποιους γενικούς κανόνες, αλλά όχι υπερβολικά αναλυτικούς, διότι μήπως δίνουμε λάθος κίνητρα στην βιομηχανία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μέγιστο όριο. Δεν μπορεί κανείς ε, να ανεβαίνει ανηφόρα 60 βαθμών ε, με τροχόσπιτο από πίσω, θεωρώντας ότι ε, αυτή είναι συνηθισμένη οδήγηση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιο σενάριο μέγιστης επιβάρυνσης, αλλά θα... Το να πούμε ακριβώς τι δοκιμές κάνουμε είναι λάθος, διότι το όχημα θα πρέπει να πληρεί κάποια όρια εκπομπών υπό κανονικές συνθήκες, υπό συνθήκε κανονικής λειτουργίας. Ε, μπορείτε λοιπόν ε, να ζητήσετε από τον ε, σύζυγό σας να δανειστείτε το αυτοκίνητο του ή και να δούμε τι απόδοση έχει ε, με οδήγηση 100 χιλιόμετρων ε, μέσα στο Βέλγιο. Εάν όλα πάνε καλά τότε έχει καλώς, εάν όχι τότε θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία. Οι αρχές ε, να αναλάβουν τη διαδικασία αυτή και να πάνε στον κατασκευαστή και να του πούνε τι τρέχει εδώ και αν το πρόβλημα υπάρχει μόνο με ένα αυτοκίνητο τότε έχει καλώς. Εάν όχι όμως θα πρέπει κάτι να γίνει. και το... Και το θέμα είναι να πάρει κανείς τρία αυτοκίνητα. Εάν το πρόβλημα υπάρχει και στα τρία, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και γι' αυτό το ΟΕΜ έχει χάσει εδώ, διότι μας είπανε «Α, ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνουμε» ε, και καταγράφουν τα στοιχεία αυτά, χωρίς όμως να τα ελέγξουν. Ευχαριστώ. Κύριε Σάλβα, έχετε γραφεί δύο φορές και ως εκπρόσωπος ε, του πολιτικού κόμματος. Εντάξει, δεν ξέρω. Αν θέλει κάποιο συνάδελφος να μιλήσει, να μην μιλήσω εγώ δύο φορέ, προφανώς. Στα ισπανικά τη μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκε που ήρθατε εδώ σήμερα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε πραγματικά. Θα σας ρωτήσω αυτό που ρώτησα και τον προηγούμενο συνάδελφο. Τώρα έχω το πλεονέκτημα ότι άκουσα τη δική του απάντηση, αλλά θέλω να ξέρω και τη δική σας γιατί υπάρχει αυτό το δίλημα στη φυσική σε όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που είναι από την ίδια την καύση. Είτε θα επικεντρωθούν ε, στην απόδοση του κινητήρα είτε θα ε, μειώσουν τα καυσαέρια αλλά θα μειωθεί και η απόδοση και η ισχύς. Ποια είναι κατά την άποψή σας η καλύτερη τεχνική λύση για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους που είναι αποκλίνοντες και αντιφατικοί μεταξύ τους. Η καλύτερη τεχνική λύση είναι ένα σύστημα καταλήτη SCR. Συμφωνώ με τον κύριο Μπόρχεστ. Εκτός από τους δύο καταλήτες που ε, μειώνουν τις, ε, τα άλλα καυσαέρια, το SCR ε, ε, στοχεύει κυρίως τα οξύδια του αζότου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η καλύτερη τεχνική λύση, αλλά πιο ενδιαφέρον είναι να δούμε σε ποιο επίπεδο ε, ε, είναι το παραδεκτό για την έκκληση αιρούμενων σωματιδίων ή οξυδίων του αζότου. Όλα αυτά είναι ε, έτσι θεωρητικά και ενημερωτικά. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την κούρσα των εξοπλισμών όπως την ονομάζω. Είναι πολύ ατυχές και λυπηρό ότι δεν υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών, καταλητών και πώς θα ελέγξουμε καλύτερα τα καυσαέρια. Όλοι το βλέπουν αυτό στην βιομηχανία των αυτοκινήτων ως ένα απαραίτητο κόστος και πάνε στον κατασκευαστή και του λένε φτιάξε κάτι ε, φτηνό που να περνάει το τεστ και το κάνανε. Και μετά αυξήθηκαν οι τιμές και είναι πιο δύσκολη η κατάσταση και έχουμε το εργοστάσιο, το χημικό και τελικά κάτω είναι ε, στη βάση του δίζελ ε, αυτοκίνητο που μπορεί να είναι ακριβό, μπορεί και όχι υπερβολικό. Μα αυτό είναι ανόητη προσέγγιση. Κανείς δεν έρχεται ε, ε με ανταμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ας πούμε, για να βρει το σωστό καταλήτη και ο καταλήτης στα περισσότερα συστήματα δεν αλλάζει. Είναι ενσωματωμένος, είναι built-in όπως ονομάζεται και το αγοράζει ο καταναλωτής γιατί είναι υποχρεωμένος να έχει ένα καταλήτη στο κινητήρα λόγω του ε, κανονισμού. Αλλά αυτά τα πράγματα χαλάνε και άμα χαλάνε δεν επισκευάζεται κιόλας. Πρέπει να βγάλεις ολόκληρο τον κινητήρα και να... Ε, ε, ε αντικαταστήσεις ένα ολόκληρο κομμάτι του άξονα ε, και ενώ θα ήταν πιο εύκολο να βγει και να κυκλωθεί κατά τα άλλα. Φυσικά δεν το κάνουν και πρέπει να χαλάσει όλη η εξάτμιση, όλος ο κινητήρας και όλα αυτά. Και δεν υπάρχει και ανταγωνισμός ε, για τους καταλήτες ε, στους προμηθευτές, γιατί είναι υπερβολική ρύθμιση και πάρα πολύ τεχνική και ο λόγος EGR, e, e ε, ε, η ανακύκλωση των καυσαερίων ε, της εξάτμισης, δεν είναι μέσα στη ρύθμιση και στον κανονισμό σου δεν είναι τιμές της πραγματικής ζωής και πώς θα το λύσει η βιομηχανία είναι δικό τους πρόβλημα. Δεν πάτε στην κοκακόλα να της πείτε τι θα βάλει μέσα στο ποτό της για να είναι καλή η γεύση. Απλώς λες απαγορεύεται να περιλαμβάνει γιατί δεν είναι ε, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, γιατί δεν είναι υγιεινό. Άρα το θέμα είναι ο κανονισμός λέτε και η ρύθμιση και όχι η καινοτομία, αν κατάλαβα καλά. Κατά την άποψή σας λοιπόν, ποια είναι η σωστή λύση για να αντιμετωπιστούν αυτά η καλή καινοτομία θα έρθει από την καλή ρύθμιση και νομοθεσία. Γιατί αν επιτρέπεται στον κόσμο να φαίνει την καλύτερη λύση υπάρχει ανταγωνισμός ε, εγκεφάλων ε, πώς θα έχουμε την καλύτερη λύση, πώς θα έχουμε τη φθηνότερη λύση. Ε, και όχι πώς θα έχουμε μια λύση που θα περνάει το τεστ. Παράδειγμα, αν μετράμε τα αυτοκίνητα επιτόπου, στο δρόμο δηλαδή και μπορούσαν όλοι ε, να συνεισφέρουν και ακτιβιστές ε, του περιβάλλοντος που ακούσατε το πρωί, τα μετράνε αυτά, αν μπορούσαν να πούνε στον κόσμο ότι κοίτα, έχω δύο αυτοκίνητα, το ένα κάνει και τα δύο 30.000, το ένα είναι πιο καθαρό και το άλλο λιγότερο καθαρό. Εμένα με νοιάζει το περιβάλλον, θα αγοράσω το πιο καθαρό. Ε, αυτή είναι η δημόσια ε, ενημέρωση. Και αυτός που φτιάχνει το δεύτερο αυτοκίνητο ή στο Δίνεκε θα είχε ένα κίνητρο για να φτιάξει πιο καθαρό αυτοκίνητο γιατί θα είχαν ανταγωνισμό. Στο παρελθόν δεν καταστήσαμε ε, πλεονέκτημα συγκριτικό το γεγονός ότι είναι καθαρό το αυτοκίνητο. Είναι κρίμα γιατί ο κόσμος πεθαίνει επειδή βγάζουν τόσα καυσαέρια τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Πώς βλέπετε το μέλλον της πετρελαιοκίνησης, είστε αισιόδοξο. Το συνδέεται με την πρόθεση της καινοτομίας. Και υπάρχει και ανησυχία γιατί είναι εκατοντάδε θέσεις και χιλιάδε θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να ανησυχούμε τι γίνεται και με αυτού του εργαζομένου, όχι μόνο για το περιβάλλον που βεβαίω και μα ανησυχεί και αυτό. Μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι και αισιόδοξοι μάλλον για τον ντίζελ. Είναι δεινόσαυρο η αυτοκινητοβιομηχανία και είναι δυσκίνητη συνήθω η δεινόσαυρη. Φυσικά θα εξακολουθεί να υπάρχει το πετρέλαιο και με περίδιο αγορά κάπου 9% σε κάποιε αγορέ στην Ευρώπη. Και ενδεχομένω ε, ε, το τελικό κέρδο για τον ιδιώτη θα είναι στο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο και λιγότερο στα πετρελοκίνητα, βενζινοκίνητα ή υβριδικά. Και το ερώτημα τώρα για τους κατασκευαστές είναι πώς το βλέπουν, ποια είναι η προοπτική, σε ποιο βάθος χρόνου, 5 χρόνια, 10 ή παραπάνω, 20. Ε, η νομοθεσία μας θα το επηρεάσει πιστεύω. Τώρα αν είναι πολύ υψηλή μπορεί να έχουμε σκοτώσει ε, και θάψει το δίζελ και το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα σε σχέση με άλλα αλλά δεν θέλουμε να καταλήξουμε σε ε, μια κατάσταση που να μην αγοράζει κανείς δίζελ ούτε στην Ασία ούτε στην Αμερική και τα δίζελ να είναι μόνο στο Παρίσι και στη Ρώμη και να γίνουν οι πόλεις αβίωτες από τον έφος επειδή έχουμε τόσα πολλά πετρελαιοκίνητα ή από την ε, άσχημη μυρωδιά, τη δυσοσμία που αφήνει το κατάλοιπο του καταλήτη. και την ε, τεχνολογία αυτή να μην την χρησιμοποιούμε απλώς επειδή τη διαθέτουμε, αλλά εκεί που μας ε, συμφέρει και βολεύει. Ε, σε μεγάλα φορτηγά, σε μηχανήματα που δεν κινούνται στους δρόμους, αλλά που είναι στατικά εγκατεστημένα κάπου οι κινητήρες. αυτό δεν σημαίνει ότι στην επόμενη γενιά θα πρέπει να έχουμε τους ίδιους κινητήρες δίζελ. Ενδεχομένω τα γιο να είναι πλήρως ηλεκτροκίνητα. Αλλά εσείς που είστε νομοθέτες, δεν σας νοιάζει πού θα γίνει η ρήπανση, αλλά να είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένο και ε, λογικό. Αν έχετε ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα στην αγορά, η ενέργεια που παράγεται για να φορτίζουν παράγεται με τρόπο που ε, να βλάπτει λιγότερο το περιβάλλον από ότι η ίδια η χρήση των αυτοκινήτων. Θα πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση και μια νομοθεσία που να κοιτάει ε, την ευρύτερη εικόνα και να αντιστρέφει το πρόβλημα. Αυτό θεωρούμε παραδεκτό στα γιοταχή. Και εκεί έχει πίεση η κοινωνία να ασκήσει. Αν θέλει κάποιος να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο για την ιδιωτική του μετακίνηση, ευχαρίστηση ή οτιδήποτε άλλο. Αν είναι μικρό το αυτοκίνητο μπορεί να είναι πιο φτηνό γιατί αν θέλετε όμως να έχετε ένα μεγάλο SUV, ε, Jeep, θα πρέπει να επενδύσετε περισσότερο στη μηχανική που έχει ένα κόστος. Που θα υπάρχει μηχανική γιατί έχει πληρωθεί το κόστος για μικρά αυτοκίνητα, για κινητήρες, ας πούμε, πλοίων ε, που δεν κυκλοφορούν στο δρόμο και τέτοια. Εσείς θέλετε να υπάρχει αυτός ο κανονισμός και αυτή η δυνατότητα. Και αν στήσετε μια καλή νομοθεσία θα γίνει. Τελευταία ερώτηση. Α, τώρα κατάλαβα γιατί είχα δύο χρονοθυρίδες. Ανησυχείτε για το πώς παράγεται η ενέργεια για τα ηλεκτροκίνητα. Και όχι πώς παράγονται οι μπαταρίες. Ε, μόνο πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια βεβαίως ανησυχώ. Και για, για το ε, βάρος ε, που κυκλοφορεί και που, και ακόμα είναι μειονεκτικό σε σχέση με την μηχανή εσωτερικής καύσης. Από πλευράς ε, μηχανικής δεν είναι τόσο καλά τα μηχανοκίνητα αυτοκίνητα, αλλά οι πολιτικοί τα έχουν βρει μεταξύ τους ότι είναι το αυτοκίνητο του μέλλοντος. Και η βιομηχανία τώρα πρέπει να πιστεί ότι είναι το μέλλον και ότι θα είναι και το έξτρα εισόδημα που χρειάζονται. Αν θέλουν να βγουν τώρα σε αυτή την αγορά και μάλιστα πολύ έντονα θα πρέπει να το ενσωματώσουμε αυτό. Η νέα νομοθεσία για τα καυσαέρια ε, στην Ευρώπη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τι είναι το αυτοκίνητο ε, και πώς ανακυκλώνεται. Ας πούμε αν είναι 200 κιλά ε, μπαταρίες λιθίου σε ένα αυτοκίνητο, τι θα γίνει μετά, πώς ανακυκλώνονται όταν χαλάνε, πώς αντικαθίστανται. Ή θα είναι ένα μεγάλο μπλοκ, θα είναι μικρά, που για να ανοίξει πρέπει να το κόψεις και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ανακυκλωθεί. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για τη νομοθεσία και για τα καυσαέρια. Γιατί αν ρυθμίσετε τώρα μόνο και νομοθετήσετε μόνο για τα βεζινοκίνητα και τα πετρελοκίνητα, τι γίνεται με την καινοτομία, με ε, την εξέλιξη και ε, με το, με το που επενδύουν. Θα πρέπει να υπάρχει καινοτομία και αν, δεν θίξετε και τα ηλεκτροκίνητα με την νομοθεσία, δεν θίξετε τον τομέα που επενδύει. Ευχαριστώ. Grazie. Ε, Ας, προσπαθούμε, προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούμε στο τι πρέπει να γίνει, στις λύσεις, πέρα από τους κύκλους ρεαλιστικούς των δοκιμών. Υπάρχουν κάποιες σκίες σε σχέση με, τα, με τους μηχανισμούς αυτούς επέμβασης και παραπλάνησης που μπορεί να είναι ύποπτη κατά κάποιο τρόπο. Εσείς τις απαντήσεις που δώσατε στην ερώτηση 6 γραπτά λέτε ότι ο ορισμός μιας τέτοιας εγκατάστασης ηλεκτρονικής από το 2007 είναι κάτι το οποίο επιτρέπει πάρα πολλά παραθυράκια. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του αγώνα που έλεγα στη λεπτομέρεια ορισμός για μηχανισμούς παραπλάνησης περιλαμβάνει ακόμα και ε, κυβότια ταχυτήτων, ε, ηλεκτρονικούς σένσορες ε, για το πώς δουλεύει το μηχάνημα αυτό. Στην ουσία αγνοεί πράγματα που έχουν οι μηχανές σήμερα και που δεν είχαν τότε. Είναι λάθος λοιπόν το να προσπαθήσει κανείς ε, να βάλει στις υπάρχουσες διατάξεις επιπλέον λεπτομερέστερες. Αν ε, κάποιος πάρει όλη την τεκμηρίωση και το λογισμικό και το ελέγξει, αυτή στιγμής θα διαπιστωστεί κάτι το αρνητικό, αν δεν είναι ακριβώς ε, αυτό που προεβλέπετε ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόστομο. Κοιτάξτε πώς τα βλέπουν τα πράγματα αυτά στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένε Πολιτείε φοβούνται τον κανονισμό, ενώ στον ευρωπαϊκό κανονισμό οι βιομηχανίες παίζουν μαζί του και αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ δεν θα ήθελα λοιπόν να βάζω ακόμα μεγαλύτερες λεπτομέρειες ή καλύτερους ορισμούς του μηχανισμού παραπλάνησης. Έχει κανείς την τεχνική τεκμηρίωση, πρέπει να δώσει στοιχεία, πρέπει να δώσει πηγαίους κωδικούς και στο τέλος το εξετάζουμε το σύνολο αυτό, το υπογράφουμε βεβαιώνοντας ότι λειτουργεί όπως προβλέπεται. Και αν δεν συμβαίνει αυτό τότε θα πληρώνει κανείς 500 ευρώ πρόστιμο αν αυτοκίνητο που βγάζει στην αγορά. Πάντα σε σχέση με το τι μένει να γίνει, λέει ο κύριος Παουλούτσι, στην ερώτηση 10. Λέτε ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε ότι η πνευματική ε, ιδιοκτησία ε, να είναι εμπόδιο στη δυνατότητά μας να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Τι είναι αυτές οι επιλογές που πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Πολύ καλή ερώτησή σας, σας ευχαριστώ για αυτήν. Ε, η νομοθεσία για την πνευματική διοκτησία ε, έχει εφευρεθεί για να επιτρέπεται κάποιοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφευρέσεις των άλλων. Κανένας δεν κυκλοφορεί αυτοκίνητα τα οποία να παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία. Και νομίζω ότι από αυτό οι άνθρωποι κερδίζουν. Όταν χρησιμοποιείται μία μέθοδος τους που έχουν δικαιώματα κτλ. Το σύστημα λοιπόν αυτό των ευρεσιτεχνιών είναι παλαιό και είναι μια λύση στα προβλήματά μας και ο κόσμος άρχισε να αποκρύβει το λογισμικό γιατί μπορεί να το κάνει ε, δυστυχώς. Μόνο και μόνο γιατί μπορεί να το κάνει. Πρέπει να σταματήσουμε το μπορεί να κάνει. Λοιπόν, πόσο μπορούμε να παρέμβουμε εδώ. Τώρα, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας τρόπος οι ρυθμιστικές αρχές να τα καλύψουν όλα μπορεί να ζητηθεί από ανθρώπους στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης τύπου να ε, αναλύεται σωστά φυσικά το σύστημα αυτό στο σύνολό του μαζί με τους πιθανούς μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμεύουν για απόκρυψη, για παραπλάνηση. Θα πρέπει λοιπόν από τη μία η βιομηχανία να προστατεύει τα δικαιώματά της τα οποία χρησιμοποιεί και από την άλλη η πολιτεία να διαβεβαιεί ότι οι νόμοι γίνονται σεβαστοί, οι ρυθμίσεις γίνονται επίσης σεβαστές. Και στην ουσία βλέπουμε ότι τα συστήματα ελέγχου και οι επιφάνειες εργασίας ελέγχου και τα λοιπά έχουν αποτύχει. Είτε δεν πήραν είδηση οπότε είναι ανίκανοι, είτε το είδαν και δεν μίλησαν, κάτι το οποίο είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια διαφορετική λύση. Εσείς σαν ρυθμιστική αρχή, σαν ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, σαν κυβερνήσεις βρείτε μια λύση ή ενημερώστε το κοινό και χρησιμοποιήστε ακριβώς ε, τις ε, δυνατότητες που δίδει η κοινωνία των πολιτών. Αν δώσετε τους πηγαίους κωδικούς στην Greenpeace θα βοηθήσει χωρίς να επηρεαστούν τα συμφέροντα των ε, προμηθευτών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Χένκελ, ευχαριστώ πολύ για το χαρακτηρισμό που ε, απευθύνεται σε αυτοκινητοβιομηχανία με την οποία, την οποία διαφωνώ απολύτως τους χαρακτηρίσατε δεινοσαύρους. Θυμίζω ότι 65 εκατομμύρια χρόνια ζούσαν οι δεινόσαυροι σε αυτό το πλανήτη, πάρα πολύ περισσότερο από ότι ε, ο άνθρωπος μέχρι σήμερα. Επίσης δεν πιστεύω ότι είναι σωστή η σύγκριση με την βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου έχω ζήσει μια ζωή. Έχουν ευθυνήνει πολλοί υπολογιστές, αλλά εμείς ως καταναλωτές δίνουμε ένα σωρό λεφτά στην Apple, στη Microsoft, την Deutsche Telekom και πάει λέγοντας. Δεν νομίζω ότι είναι λογικός αυτός ο χαρακτηρισμός ότι είναι υποπιστοδρομική δεινόσαυρη αυτοκινητοβιομηχανία. Επίσης, ε, πέσατε στην παγίδα να γενικεύσετε το θέμα, το πρόβλημα της Volkswagen. Είπατε και πάλι ότι Ε, ότι το γενικεύσατε για όλους τους Ευρωπαίους, ότι είπατε ότι οι Ευρωπαίοι παίζουν παιχνίδια. Εγώ φίλω αυτό να το αποκρούσω και να το αντικρούσω. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε στηρούν τους κανόνες. Θαυμαστά αυτό που μας λέτε ως δηλώσεις. Να τα ξανασυζητήσουμε όταν θα συζητάμε το TTIP ε, μία από αυτές τις μέρες. Μία ερώτηση έχω και μοναδική και είναι εξή. Δεν θα ήταν καλή ιδέα κατά την άποψή σας να προσθεθεί αυτό το θέμα των κανόνων και των προδιαγραφών στις διαπραγματεύσεις για το TTIP. Απάντησε. Ε, λάθος με παραθέσατε εγώ, είπα ότι αυτοκίνητο βιομηχανία φοβάται ε, τις ε, προδιαγραφές των ΗΠΑ και παίζει παιχνίδια με τις ευρωπαϊκές για να το διορθώσουμε αυτό. Δεν έχω ιδέα για το TTIP. Εγώ είμαι μηχανικός, είμαι σύμβουλος σε πολλούς τομείς, αλλά όχι στο συγκεκριμένο. Δεν έχω ιδέα ε, για το TTIP ούτε τι περιλαμβάνει, ούτε αν έχει νόημα να προσθεθεί το συγκεκριμένο θέμα ή όχι. Ο κύριος Γερμπράντη. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία στο ερωτηματολόγιο τα οποία δεν θίξαμε. Έχω όμως μια άλλη ερώτηση. Έχετε εξετάσει αναλυτικά το λογισμικό και έχετε εργαστεί στο, στην BMW στο παρελθόν. Γνωρίζετε ότι η έγκριση τύπου βασίζεται στο λεγόμενο χρυσό αυτοκίνητο, το οποίο έχει κάποια σχέση με το αυτοκίνητο που θα απολυθεί μετά από ένα μήνα στους καταναλωτές, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφορές. Εξετάσατε ποτέ την διαφορά ανάμεσα στο χρυσό αυτοκίνητο και το τελικό αυτοκίνητο που ε, πολίθηκε. Μάλλον συμμετείχατε στις διαφορές αυτές. Όχι, όχι, είχα να κάνω με το λογισμικό και με την επιστοποίηση των αυτοκινήτων. Δεν είχα σχέση με αυτό που λέτε. Δεν γνωρίζετε πόσο σημαντικές είναι οι διαφορές ανάμεσα στο χρυσό αυτοκίνητο και το τελικό προϊόν. Όχι, δεν είδα να υπάρχουν. Όπως είπε ήδη ο κύριος Μπόρκεστ, δεν υπάρχει μόνο μία εκδοχή του λογισμικού σε ένα μοντέλο. Δεκάδες διαφορετικά λογισμικά υπάρχουν, μερικά για να διορθώσουν λάθη, μερικά για να βελτιώσουν την απόδοση, μερικά ε, για ε, να διατηρηθεί η τυποποίηση ανάμεσα στο παλιό και στο νέο μοντέλο. Ε, κάποιο λογισμικό έχει να κάνει με την συντήρηση του αυτοκινήτου. δεν είδα αυτό που υποβάλλεται κατά την έγκριση τύπου να είναι σκεμμένα διαφορετικό από την εκδοχή που ε, τοποθετείται στα αυτοκίνητα που θα απολυθούν τελικά. Αυτό που βλέπουμε είναι διαφορές ανάλογα με τις ε, συνθήκες, αλλά γενικά υποτιμάται η διαδικασία ανάπτυξης ε, του λογισμικού. βλέπουμε συχνά ότι πρέπει να φορτίσει κανείς σε λογισμικό επί 3-6 ώρες. Ε, ο κύριος Κερβάντη, ναι, αλλά βλέπουμε ότι συχνά η έγκριση τύπου βασίζεται στο χρυσό αυτοκίνητο. Αλλάζουν λοιπόν πολλά μετά από αυτό. Ε, ο κύριος Λάνιε, νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι παρουσιάζουμε αυτό το αυτοκίνητο, το εγκρίνουμε και μετά δεν το ξανακοιτάμε. Ε, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα αυτή. Οι Αμερικανοί ε, το κάνουν επιλέγοντας ε, τα αυτοκίνητα που θα ελέγξουν. Έτσι το κάνει η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα πρότεινα να ανοίξουμε τη δυνατότητα αυτή και για άλλους ενδιαφερομένους στην αγορά, ομάδες ακτιβιστών, ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Και προφανώς ε, και στους ε, τοπικούς επιθεωρητές. Έτσι λοιπόν συγκεντρώνει κανείς πολύ περισσότερα δεδομένα. Εάν δηλαδή δημοσιεύσει κανείς τα δεδομένα σε ένα μορφότυπο που να μπορεί να διαβάσει ο κόσμο. Ε, τότε από μόνη τη αναπτυχθεί αυτή η δυναμική, διότι υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των ανθρώπων. Εάν αγοράσουν ένα αυτοκίνητο που στοιχίζει 45.000 ευρώ, ε, θα θέλουν να τα γνωρίζουν αυτά. Ωραία, ευχαριστώ. Και η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με την εμπειρογνωμοσύνη. Έχετε την ε, εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή οι δημόσιες αρχές έχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για να κάνουν αυτά που πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν. ή πρέπει να βασίζονται στην κοινωνία των πολιτών, όπως ήδη αναφέρατε. Είναι τεράστιο το εύρος ε, της τεχνογνωσίας ε, στις διάφορες ε, ρυθμιστικές αρχές. Έχω συνεργαστεί με κάποιες από αυτές το τελευταιο εξαμηνο εξάμηνο-επτάμηνο. Υπάρχουν άνθρωποι με πάρα πολλές γνώσεις υπό μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν άλλοι με πλήρη άγνοια της τεχνολογίας σε, σε άλλη γειτονική χώρα της προηγουμένης. Προφανώς υπάρχουν οι, οι ιστορικοί λόγοι για κάτι τέτοιο. Κάποιοι έχουν πρόσβαση σε καλά πανεπιστήμια, άλλοι όχι. Δεν νομίζω ότι είναι ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών να είναι εμπειρογνώμονες απαραίτητα, αλλά πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη και να διασφαλίζουν την επιβολή του νόμου. Δεν μπορεί κανείς να είναι εμπειρογνώμονα σε όλους τους τομείς που ρυθμίζει. Δεν θα ξεκινούσα λοιπόν καν μια τέτοια προσπάθεια. Κατά τη σύγκριση της ε, των διαφόρων προμηθευτών. Θα διαπιστώσουμε ότι κάποιοι δεν είναι τόσο καλοί, που προφανώς είναι αυτοί που δεν ε, έχουν βρει τις ε, καλές ε, συσκευές αναστολής. Κυρία Κονέτσινα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Λάγκε για την ειλικρίνεια στις απαντήσεις τους ε, και ε, ε, γραπτός επίσης ήταν πολύ ειλικρινής, δεν είναι καθημερινή πρακτική αυτή. Θέλω να ρωτήσω και εγώ κάτι που ρώτησε ο κύριος Γκεμπράντη. Αφήσατε να εννοηθεί ότι οι ρυθμιστικές αρχές, το γράψατε και στις απαντήσεις σας, ότι δεν πληρούν τα προσόντα να συνεχίσουν να ελέγχουν αυτόν τον κλάδο. Και είπατε ότι δεν έχουν την πραγματογνωμοσύνη. Αυτό φταίει. Ή μήπως υπάρχουν ε, ε, συμφέροντα, ε, χειραγωγούνται από διαφόρους που εκείνοι έχουν συμφέροντα. ναι. Υπάρχουν δύο πλευρές εδώ που πρέπει να τονίσουμε. Από τη μία, ο νέος ευρωπαϊκός κύκλος είναι κακή νομοθεσία και ήταν κακή ήδη από την αρχή. Και είναι κακό επίσης δύο φορές το ότι ισχύει τόσο πολύ καιρό και νομίζω ότι οι σωστοί στα πλαίσια των ρυθμιστικών αρχών γνωρίζουν ότι δεν είναι ικανοποιητικό. Οι συζητήσεις γίνονται εδώ και 10-12 χρόνια και ξέρετε πως πάνε αυτά στην πολιτική. Έχει ενδιαφέρον να συζητάει κανείς τα πράγματα επί μακρόν και όχι να αναζητεί ένα κοινό τρόπο και να κάνει τις αλλαγές ένα-δυο χρόνια είναι δεινόσαυροι αλλά παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα κινητικοί και κάθε τόσο βγάζουν καινούργια αυτοκίνητα και ρίχνουν στις αγορές. Οπότε δεν μπορεί κανείς να έχει έναν κανονισμό ο οποίος να είναι αποτελεσματικός για 20 ολόκληρα χρόνια. Οι ρυθμιστές λοιπόν, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ξυπνήσει το ότι υπάρχει αυτό το σύστημα δείχνει ότι προσπαθείτε να αλλάξετε την κατάσταση, βλέπετε ότι το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε πολιτικό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν, είμαι αισιόδοξο ότι στις εκθέσεις σας θα υπάρχουν εξαιρετικές προτάσεις που θα βελτιώνουν το διακανονιστικό πλαίσιο και δείτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σαν παράδειγμα. Αυτό είναι το μέλλον υποτίθεται θα πρέπει να τα ρυθμίσετε με έξυπνο τρόπο. Έχετε αυτοκίνητα που λέγουν ότι έχουν ε, ε αυτάρκεια για 160 χιλιόμετρα, ακτίνα δηλαδή, ενώ οι κατασκευαστές λένε ότι κοιτάξτε αυτός είναι ο επίσημος αριθμός, ίσως να είναι και 130. Και αν ένα παγωμένο πρωινό στη Γερμανία με μείον 10 βάλετε και το καλοριφέρ, βάζετε και το GPS και το ραδιόφωνο, τότε δεν ξεπερνάτε τα 75 χιλιόμετρα και ξαφνικά μένει το αυτοκίνητο από μπαταρία. Λοιπόν πρέπει να τα ρυθμίσετε αυτά, υπάρχει ανάγκη. Αν πουλεί κανείς ένα αυτοκίνητο που λέει ότι μπορεί να καλύψει 170 χιλιόμετρα, ίσως εν πάση περιπτώσει σε 10 χρόνια να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα. Δεν εμπιστεύεται ο κόσμος τις ε, υποσχέσεις των κατασκευαστών σε σχέση με την εμβέλεια. Δίνουν ένα μέγιστο το οποίο δεν είναι επιτεύξιμο παρά μόνο αν το σπρώχνεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την απάντηση. Έλλη μια ερώτηση. Ε, σε μια από τις απαντήσεις σας, σωστά είπατε, ότι υπάρχει ένας κύκλος σιωπής ε, και τη χειραγώγηση για τα καυσαέρια. Εμείς λέμε τώρα ότι αυτές οι εκπομπές χειραγωγούνται εδώ και 10 χρόνια. Και ήταν κοινό μυστικό. Και το σύστημα ήταν πάρα πολύ περίπλοκο και άχρηστα πολύπλοκο από το σχεδιασμό του. Αυτό που με ενοχλεί εμένα και με προβληματίζει είναι πώς και δεν υπήρχε κανένας καταγγέλων whistleblower από ορισμένους που απολύθηκαν ενδεχομένω από αυτές τις εταιρείες. Πώς το βλέπετε, γιατί αυτή ομερτά. Φοβούνται οι υπάλληλοι. Περίεργο, δεν άνοιξε κανείς το στόμα του 10 χρόνια τώρα. Ναι, δεν άνοιξε το στόμα του 10 χρόνια, διότι τουλάχιστον τόσο χρειάστηκε και στη Volkswagen. Η Mitsubishi βγήκε και είπε 30 χρόνια κάνει τέτοια πράγματα με τις δοκιμές για τις εκπομπές καυσαερίων και ε, την κατανάλωση. Ευκαιρίες υπήρχαν, αλλά όπως σας είπα και εισαγωγικά, ο κόσμος όταν ανοίγει το στόμα του θα πρέπει να αισθάνεται μια σιγουριά. Γιατί όταν είναι μια οργάνωση, ένας οργανισμός με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που ξέρουν ε, ότι ε, υπάρχει μια εξαπάτηση και βγεις εσύ και το πίστος, τότε εσύ είσαι το μαύρο πρόβατο. Αυτό δεν θα ξαναβρει δουλειά στην αυτοκινητοβιομηχανία, ούτε στου προμηθευτέ, ούτε πουθενά. Κάπου πρέπει να έχει ένα μέλλον αυτό για να ανοίξει το στόμα του, να προστατεύεται και νομικά και να αποζημιωθεί για το διαφυγόν κέρδο. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό για τα καυσαέρια μόνο από την αυτοκινητοβιομηχανία. Ας πούμε κάποιος που καταγγέλει οποιαδήποτε θέματα ε, περιβαλλοντικά. Αν επιβεβαιωθεί, αποζημιώνεται για την απώλεια εισοδήματος και το διαφυγόν κέρδος. Και μπορεί να πάρει και μπόνους επιπλέον. Πέρα από το πρόστιμο που θα επιβληθεί, στον, θα πάρει ένα ποσοστό. Έλα, δεν είναι μόνο αυτό. Ε, χρειάζεται κάποια βεβαιότητα και κάτι άλλο να πω. Ο κόσμος θα πρέπει να πηγαίνει σε εταιρείε και να ανακοινεί το θέμα εσωτερικά. Ε, και αν δεν λειτουργεί στο εσωτερικό της εταιρεία, μπορεί να χρειαστεί ένας προστατευμένος όμως ε, τρόπος δημόσιος να καταγγείλει αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ όλα όσα είπατε σχετικά με τη βελτίωση του συστήματος. Η δουλειά μας όμως ε, στην ε, έρευνα αυτή είναι ε, η λογοδοσία από πλευρά των αρχών. Ας μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Θα σας δείξω μια διαφάνεια. Αν κατάλαβα σωστά την ομιλία σας με τον Φίλιπ Τόμκε, από την οποία προέρχεται αυτή η διαφάνεια, οι τρεις κάτω γραμμές δείχνουν, η μεσαία δείχνει ε, τις αποστάσεις που έχουν οδηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι άλλες δύο γραμμές δείχνουν ένα ε, στενό διάδρομο στον οποίο ε, βλέπουμε τα όρια από τα οποία μπορούν, κατά τα οποία μπορούν να αποκλίνουν. Ναι, αυτό είναι αυτό που βρήκε ο Φίλιπ σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος. Η λευκή γραμμή λοιπόν ε, δείχνει την απόσταση στο χρόνο που δίνει ο Φίλιπ. 1200 δευτερόλεπτα. Εάν λοιπόν παραμείνει εντός αυτής της ζώνης, ε, το αυτοκίνητο ε, λειτουργεί με καθαρό τρόπο. Εάν ξεφύγει από αυτόν, ε, τότε δεν λειτουργεί με καθαρό τρόπο και μπορεί να έχει 30 φορές τις εκπομπές που έχει εντός του διαδρόμου. Αυτό λοιπόν είναι νόμο. Όχι, η Volkswagen συγκεκριμένα ο κύριος Όραν ε, μπροστά σε ε, Αμερικανικό Ρυθμιστικό Συμβούλιο παραδέχτηκε τη χρήση συστήματος αναστολής ε, και είπε ότι δεν προστατεύει τη μηχανή, απλά στόχο έχει την απάτη. Δεδομένης της πείρας σας, πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να αναπτύξει λογισμικό και να το ενσωματώσει σε αυτοκίνητο χωρίς να το γνωρίζουν οι ανώτεροί του. Ή μπορεί να το κάνει αυτό ο κατασκευαστή του ECU χωρί να το γνωρίζει ο κατασκευαστή του αυτοκινήτου. Όχι, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η BOS ε, να ε, θέσει σε λειτουργία τις ε, γραμμές αυτές. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Volkswagen. Υπάρχει η ανάπτυξη του λογισμικού και υπάρχει η ρύθμιση του η οποία πραγματοποιείται στην Volkswagen σε αντίθεση με την ανάπτυξη που γίνεται στην Bosch. Δηλαδή η Bosch αναπτύσσει το λογισμικό, η Volkswagen το ρυθμίζει. Και ουσιαστικά μπορούν να αφαιρέσουν το σύστημα αναστολής ε, σβήνοντας τις γραμμές αυτές ε, Εσείς και ο κύριος Ντόμ και βρήκατε ανάλογα πιστικά στοιχεία σε άλλα αυτοκίνητα άλλων ε, κατασκευαστών. Ο Φίλιξ συνεργάστηκε με ομάδα δημοσιογράφων ε, από το NDR και το Spiegel και βρήκε σύστημα αναστολής σε αυτοκίνητα της Opel. Πιθανότατα υπάρχουν ε, πολλές ε, συσκευές αναστολής ε, που σχετίζονται με το παράθυρο των θερμοκρασιών, με το φάσμα των θερμοκρασιών. Η κανονική χρήση, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είναι σε θερμοκρασίες ε, κάτω των 70 ε, βαθμών. Αυτό στην ε, Γερμανία δεν είναι δυνατόν, στη Σκανδιναβία ίσως ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο. Είναι τέτοιος που ουσιαστικά μειώνεται ή σβήνει το σύστημα ε, του καταλήτη. Το θέμα δεν είναι μόνο η νομοθετική ρύθμιση που δεν είναι πολύ καλή εδώ. Ε, υπάρχει και το πνεύμα του νόμου το οποίο σαφώς παραβιάζεται εδώ πέρα και μάλλον γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσετε λογοδοσία. Και μια τελική ερώτηση, δεδομένου ότι η Εθνική Αρχή έχει εγκρίνει το αυτοκίνητο αυτό με αυτό το σύστημα αναστολής και εφόσον ε, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τον κανονισμό υποκανονικές συνθήκες, πιστεύετε ότι κάνουν τη δουλειά τους όσον αφορά την επιβολή του νόμου. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας. Ε, ε, διάβασα την έκθεση. Ε, ανέκδοτο είναι. Λυπάμαι που το λέω. Έχει γραφεί η έκθεση αυτή με στόχο να αθωώσει ουσιαστικά το σύνολο της ευρωπαϊκής αυτοκίνητοβιομηχανίας ή μέρος της. Ε, τώρα υπάρχουν κάποιες ε, διαμάχες με την ε, Ιταλική βιομηχανία διότι προσκλήθηκε να εξηγήσει στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία πώς λειτουργεί το σύστημα αναστολής τους, αλλά ουσιαστικά σβήνει μετά από ένα χρονικό διάστημα και προσκλήθηκαν και δεν εμφανίστηκαν. Και αυτή ήταν η μόνη φορά που από ό,τι γνωρίζω το, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία είπε ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, πρέπει να έρθετε και να μας εξηγήσετε το θέμα αυτό. Αλλά εγώ ως μηχανικός διαβάζοντας ε, την έκθεση γελούσα. Ε, Υπάρχουν εδώ στοιχεία που δείχνουν υπερβολικέ εκπομπέ. Ε, ζητήθηκε από τον ε, κατασκευαστή να το σχολιάσει αυτό και αυτός είπε ότι, α, μάλλον μετρήσατε λάθος Οπότε η υπηρεσία λέει ότι, α, μάλλον εμεί κάναμε λάθος οπότε αφαιρούμε το στοιχείο αυτό από την έκθεση. Grazie per le sue risposte. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρόσκληση αυτή που κάνατε και εσείς και ο πρωινός ομιλητής αναφερθήκατε και στα Ιταλικά αυτοκίνητα και που έχουν και αυτά τη δυνατότητα να σταματούν τη λειτουργία του software δύο λεπτά αμέσως μετά το τέλος του κύκλου δοκιμών. Θα θέλαμε από τις Ιταλικές αρχές να γνωρίζουμε αν έγιναν κάποιες έρευνες και αν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Γιατί μέχρι τώρα σιωπούν. Μία άλλη ερώτηση θα ήθελα να κάνω σχετικά με τους λεγόμενους παράγοντες συμβατότητας ή συμμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη το ότι υπάρχουν οι τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασκευαστές γνωρίζουν από το 2007 ότι θα όφυλαν να σεβαστούν συγκεκριμένα όρια από το 2014 ή 2015 για όλα τα αυτοκίνητα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι κατασκευαστές όλοι έτυχαν χρηματοδότησης και κινήτρων για να πετύχουν την χρήση τεχνολογιών μείωσης των νόξ και γενικά των ουσιών που μολύνουν, εις βάρος τα κίνητρα αυτά βέβαια των καταναλωτών, κόστισαν στους καταναλωτές τους ίδιους, εσείς πιστεύετε ότι η παραδοχή ότι η περίοδος αυτή που προβλέπεται για την εφαρμογή του νέου κύκλου είναι πάρα πολύ γενιόδορη και όχι ιδιαίτερα εύθετη και στην ουσία θα επιτρέψει να μην αποσυρθούν τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη σήμερα. Κάτι το οποίο ουσιαστικά λέει ο ίδιος ο κανονισμός ότι θα έπρεπε να γίνει ότι θα πρέπει να αποσυρθεί η έγκριση τύπου των αυτοκινήτων τα οποία δεν σέβονται τον κανονισμό. Νομίζω ότι το θέμα αυτό έχει συζητηθεί εδώ και αρκετό καιρό και ήταν μια δίκαιη αντιμετώπιση των κατασκευαστών. Να τους πούμε ότι σε 5-10 χρόνια θα το πετύχετε και αυτά είναι τα στάδια μέχρι τότε. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, είναι θέμα εμπιστοσύνης. Θα πρέπει οι ρυθμιστικές αρχές να είναι αξιόπιστες. Εφόσον λοιπόν τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι είχαμε, θα εμείνουμε σε αυτό. Το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει. Δεν θα ήταν ιδιαίτερα δίκαιο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου να πληρώσει το τίμημα της εισαγωγικά ατιμίας του κατασκευαστή του. Δεν θα αποσυρθούν λοιπόν όλα τα αυτοκίνητα. Ο κύριος Μπόρχες μίλησε και για την εκ των υστέρων εγκατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Το θέμα είναι ότι τα αυτοκίνητα δεν έχουν διάρκεια ζωής μεγάλη πια. Άντε δέκα το πολύ ενώ παλιά ήταν 15 ή 20. Τώρα υπάρχουν περισσότερο ηλεκτρονικά, είναι δύσκολο να επισκευαστούν, οπότε οικονομικά δεν είναι βιώσιμο να κρατά κανείς αυτά τα αυτοκίνητα σε κυκλοφορία. Συνεπώς λοιπόν το πρόβλημα αυτό θα λυθεί μόνο του σιγά σιγά. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι να καταλήξουμε σε ρυθμίσεις βελτιωμένες όπως είπαμε, αμέσως μετά ή γρήγορα μάλλον μετά από την θέση σε λειτουργία του νέου κανονισμού. Από το 2017 θα έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα λέγει τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξετε το σύστημα σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει τα στοιχεία του κύκλου δοκιμών να ανταποκρίνονται σε ένα πραγματικό κύκλο οδήγησης και πόσες παραβιάσεις μπορούμε να δεχτούμε σαν στατιστικό λάθος. Αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε το σύστημα. Το RDA λοιπόν είναι ένα καλό σύστημα, συνεχιστεί, να λειτουργεί, συνεχιστεί η λειτουργία του, περιμένοντας κάτι το οποίο ε, θα περιλαμβάνει όλα και τα υβριδικά και τα ηλεκτροκίνητα, να μην μείνουμε μόνο σε αυτά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και άλλες νέες μορφές χρήσης των οχημάτων σήμερα, όπως το car sharing. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρέφιν Φοντούν Χόνσταϊν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω. Στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα γιατί είπατε ότι ως μηχανικός δεν τα θεωρείτε τόσο καλά, αναφέρατε διάφορους λόγους, μερικούς γιατί δεν τα θεωρείτε τόσο καλά, αλλά είπατε ότι οι πολιτικοί τα προωθούν. Μάλιστα. Για μας είναι σημαντικό το θέμα εδώ όμως. 160 ή 75 ε, χιλιόμετρα, εντάξει, άλλα είναι πιο ακριβά, πιο φθηνά, οι ε, εξελίξεις τρέχουν ραγδαία, αλλά δεν το βλέπετε ως αναλλακτική λύση. Ε, ε, θα επιλέξουμε τη ρήπανση, τώρα τι θα ρηπαίνουμε, την ατμοσφαιρικό αέρα ή το νερό. Ενώ για τις μπαταρίες, τις ορευτές, αυτό το συζητάτε καθόλου ή μπα η νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ε, θα υπάρχει ανακύκλωση και ότι η ανακύκλωση ε, ανταποκρίνεται σε περιβαλλοντικές ε, προϋποθέσεις, όχι να τις στέλνουμε στην Αφρική, να τις καίνε σε τίποτα παράνομες. Αυτό δεν είναι λύση. Λύση θα πρέπει να είναι η ρύθμιση για ε, το πώς αποσύρονται, το πώς διαλύονται αυτά τα αυτοκίνητα και πώς ανακυκλώνονται. Και αυτά να ε, ε, είναι γνωστά δημοσίως. Γιατί αν υπήρχε δημόσιος έλεγχος δεν θα έστελε κανείς τις μπαταρίες να τις κάνει στην Αφρική σε συνθήκες ανεξέλεγκτες. Στο παρελθόν αυτό ήταν το πρόβλημα ότι ήταν ε, μια σιωπηρή διαδικασία μεταξύ των ε, εταιριών, των κατασκευαστών και των ενδιαφερομένων. Αλλά το κοινό δεν το ήξερα. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, δημόσια γνώση, γιατί για ποιο λόγο να τα κρύβουμε αυτά τα πράγματα αν τεχνικά υπάρχει δυνατότητα και σας είπα ότι εγώ είμαι μηχανικός και μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ εύκολη, όχι εύκολη, υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης των ε, συσσωρευτών λιθίου. Ε, βέβαια έχει και το κόστος το αυτό. Ε, ε, με την ανακύκλωση κάποιο από το κόστος καλύπτεται, πάντως η δυνατότητα να ανακυκλωθούν υπάρχει. Άρα δεν είναι και τόσο κακά τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα ή, βελτιώνονται όσο πάνε. Ε, το, πρόβλημα είναι το τεχνικό μειονέκτημα ότι κουβαλάνε 200 κιλά μπαταρίες που ζυγίζουν το ίδιο είτε είναι άδειας είτε είναι γεμάτες. Ε, ενώ όταν φουλάρεις πετρέλαιο βάζεις 50 λίτρα και όταν αδειάσει το ρεζερβουάρ δεν έχει τίποτα, δεν ζυγίζει τίποτα. Ενώ οι μπαταρίες είναι ένα βάρος που κουβαλάς γεμάτες άδειες το ίδιο. Αυτό είναι ε, ένα τεχνικό στοιχείο. Θα ήταν λιγότερο ζήτημα ε, όσο προχωράει ο χρόνος και αν αρχίσει ο κόσμος να δεν πιστεύετε ο κόσμος δεν, δεν κάνει μεγάλες αποστάσεις για τη δουλειά του. Από το πολύ 20 χιλιόμετρα πήγαινε έλα και μπορεί να χρησιμοποιεί το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Αλλά για μεγαλύτερες αποστάσεις, αν θέλει να πάει μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, δεν το εμπιστεύεται. Σου λέει και άμα μείνω από μπαταρία, τα στοιχεία δεν είναι σωστά ή δεν είναι αξιόπιστα, δεν το εμπιστεύομαι. Κύριε Σερτούκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάνε. για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Ε, θα ήθελα να επανέλθω στην ε, διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού. Ε, αναφέρεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Αλλά ποιος τη βλέπει την τεκμηρίωση αυτή. Ποιος την ε, διατηρεί, πόσα αντίγραφα υπάρχουν. Υπάρχει η σχετική τεκμηρίωση σε αυτόν που αναπτύσσει ε, το λογισμικό, στην Πόση για παράδειγμα η οποία δεν, απευθύνεται, δεν είναι απαραίτητα προσβάσιμη από τον πελάτη, την Volkswagen δηλαδή. Και υπάρχει και η εκδοχή που δίδεται στον πελάτη. όπου υπάρχει μια δημόσια λίστα των τροποποιήσεων που έχουν γίνει. Ενδιαφέρον για τις ρυθμιστικές αρχές. Είναι οι τροποποιήσεις που εσκεμένα έχουν γίνει. Όσον αφορά, για παράδειγμα, ε, τα συστήματα αναστολής, τα οποία ε, δεν βρίσκονται εκεί τυχαία. Και ο Φέλιξ απέδειξε ότι υπήρξε και συντήρηση των συστημάτων αναστολής, υπήρξαν διορθώσεις, ε, διότι υπήρχαν λάθη στην αρχή. Ε, φαίνεται δηλαδή ότι είναι ένα προϊόν το οποίο συντηρούν κιόλα. Όλοι λοιπόν οι διαπιστευμένοι οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτό. Θα γνωρίζετε ότι σε κάποιους ε, κατασκευαστές ε, υπήρξε κατάσχεση υλικού από τις γαλλικές αρχές, ε, τις γερμανικές, για τις γαλλικές δεν ξέρω, που απέκτησαν αντίγραφα του λογισμικού αυτού και διαπίστωσαν ποιος έχει αναπτύξει το σύστημα, ποιοι είχαν πρόσβαση, ποιος έχει υπογράψει τα σχετικά έγγραφα κλπ. Όπως όμως είπα κατά την ε, εισαγωγή μου, το να τιμωρηθούν αυτοί είναι η μισή δουλειά. Το θέμα είναι κατά πόσο το γνωρίζουν αυτό οι διευθυντές, διότι ε, ο κόσμος ε, δεν εξαπατά επειδή θέλουν, αλλά επειδή πιέζονται από πάνω και πρέπει να πληρώσουν τον νίκη και έχουν και δύο παιδιά. Αυτό που μόλις περιγράψατε δεν θα πρέπει να απασχολήσει το κοινό κέντρο ερευνών. Δυστυχώς ε, δεν γνωρίζω τόσο καλά ε, τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να σας δώσω μια ε, εμπεριστατωμένη απάντηση. Αλλά το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε σωστή νομοθεσία που να αντέξει και στο μέλλον, θα πρέπει να ε, συζητιέται και με εμπειρογνώμονες. Ε, το αν αυτό θα το κάνει ε, το Κοινό Κέντρο Ερευνών ή κάποιος άλλος, αυτό θα πρέπει εσείς να το αποφασίσετε. Εγώ δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να σας απαντήσω. Ο κύριος Σούλσε. Κύριε Λάγκε, σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας λέτε. Έχω πολλές ερωτήσεις Προηγουμένως, πριν από λίγα λεπτά, μιλήσατε για την εξιντόπερν και είπατε ότι αυτό, όταν τα είδατε βάλετε τα γέλια ή εξεπλάγετε κάτι τέτοιο. Να γελάσουμε κι εμείς. Θα τα μοιραστείτε αυτά μαζί μας. Δεν λέω να τα πείτε τώρα, γραπτός θα μας τα διαβεβάσετε. Ποια σημεία βρίσκεται τόσο ενδιαφέροντα ή τόσο αστεία γιατί θα μας ενδιαφέρει και εμάς ως βουλευτές να έχουμε άποψη για αυτή την έκθεση. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα δεν θέλω να ανοίξω έναν ανταγωνισμό, τι λέει ο ένας εμπειρογνώμων και τι λέει ο άλλο. Να σας πω δύο πράγματα που είναι στραβά. Αυτή η διαδικασία δεν έγινε δημόσια. Δηλαδή έγιναν κάποιες δοκιμές, οι δοκιμές συζητήθηκαν με τους κατασκευαστές και μετά το αποτέλεσμα και ένα τμήμα της ε, ε, αξιολόγησης βγήκαν προς τα έξω. Αλλά ούτε τα πρακτικά της συνεδρίασης, ούτε ε, οι χοντρικές τιμές των μετρήσεων, οι ακατέργαστες δεν βγήκαν στη δημοσιότητα. Αυτό αφήνει μια πικρή γεύση. Όταν βλέπεις ένα αποτέλεσμα που δεν σου κάνει, το ξαναμετράς ως μηχανικός και μετράς τρεις φορές ε, και όταν δεν σου κάνει το αποτέλεσμα, δεν φταίει το αποτέλεσμα, αυτέ εσύ που κάτι έχει πάει στραβά και ψάχνεις. Ε, γενικά ήταν η χρονική πίεση, κάνανε διάφορα σενάρια, πάρα πολλά αυτοκίνητα, αλλά αυτό δεν είναι δήλωση. Ε, η... Ε... να πει ότι α, μετρήσατε λάθος. Τώρα να μην πω σε λεπτομέρειες για τα φίλτρα των νεωρούμενων σωματιδίων. Υπάρχουν ε, τα ηλεκτρονικά στοιχεία για τις, διά, τις on board, όπως λέγονται ε, αυτά, και όταν είσαι μηχανικός και, και κάνεις μετρήσεις και δοκιμές, καταλαβαίνεις τι αποτέλεσμα βγάζεις και δεν χρειάζεται μια ρυθμιστική αρχή. Εντάξει, ε, τώρα μακρηγορήσατε και μου φάγατε χρόνο με την απάντησή σας. Έχω και άλλο χρόνο και θα παραμείνω. Εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, και στην Επιτροπή μας αυτά που λέτε βγαίνουν και προς τα έξω. Και αν κάνετε τέτοιες δηλώσεις, επειδή μεταδίδεται η συνεδρίαση, αμφισβητείτε την έκθεση αυτή και θα σας παρακαλούσα γραπτός να τοποθετηθείτε και σε λεπτομέρειες να μας εξηγήσετε ποια από τα σημεία αυτά για ποιους λόγους ε, δεν είναι σωστά. Και είναι και τόσα αστεία που σας κάνω να γελάτε και να κάνετε τέτοιες δηλώσεις. Γραπτός. Ε, θα απαντήσετε ή όχι, θα μου πείτε ότι δεν θα το κάνετε. Μπορείτε να μου το αναθέσετε αν θέλετε. Εγώ είμαι σύμβουλο και είμαι και προς ενοικίαση. Ε, ε, αμείβομαι γι' αυτό το λόγο. Αλλά δεν ε, μπαίνω στο ρόλο του ανταγωνισμού των εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή Ντόμπριν είχε μια εντολή για το Υπουργείο να προετοιμάσει μια βάση πληροφοριών. Κάνανε μια σειρά δοκιμών που είναι καλές δοκιμές και μαθαίνεις πολλά, αλλά στην αξιολόγηση λίγο κάναν κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου δεν είναι καλή μηχανολογική δουλειά, μηχανική. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, αλλά να σας κάνω εγώ τώρα την αντιέκθεση, δεν θα το κάνω. Ε, ωραία. Τώρα για λεπτομέρειες, γραπτός. Λέτε να το τώρα θέσουμε, δηλαδή επαμοιβή εννοείται. Μισή σελίδα μπορώ να σας γράψω για το που έβαλα τα γυαλιά ε, ε, και δωρεάν. Ε, με χαρά. Αλλά η κανονική μέθοδος θα ήταν να κοιτάξουμε από ευρωπαϊκής πλευράς τι έγινε ε, σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων. Η κυρία Σεγκολέν Ρουαγιάλ, υπουργό Περιβάλλοντος της Γαλλίας, βγήκε στον τύπο την επομένη ε, του, της έρευνας ε, στα γαλλικά εργοστάσια και είπε ότι δεν έχουν τέτοιες συσκευές οι Γάλλοι. Πολύ γρήγορα το βρήκαν. Ο κύριος Ντόμπριν, ο Γερμανός Υπουργός, ε, είπε ότι όλα ήταν καλά γιατί τα ξεπλύνανε και μετά ήρθε ο Φέληξ και είπε από 17 βαθμούς Κελσίου μέχρι 35 πάει εντάξει, αλλά παραπάνω παρακάτω όχι. Ε, αλλά επέλεξαν θερμοκρασίες 20 με 30 βαθμούς που ξέρανε ότι είναι εντός αυτή τη θηρίδας. Όταν μετράς κάτι ε, και δεν το βρίσκεις, τότε δεν έχεις ε, ενδεχομένω τα σωστά στοιχεία ούτε τη σωστή εντολή. Πόση ώρα θα μιλάτε κύριε Σόλτσα, ο κύριος Ζωρίνιο. Θα μιλήσω πορτογαλικά να σας συγχαρώ για τις δραστηριότητε σας, για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα για να εντοπίσετε αυτές τις πρακτικές εξαπάτησης. Σας ευχαριστώ επίσης και για τις εξαιρετικές σας απαντήσεις. Μας είπατε ότι είστε μηχανικός και ειδικό σε θέματα στρατηγικής. Ε, αν σας ζητήσουμε μία συμβουλή αν μια επιχείρηση θέλει να κάνει μια επένδυση για το μέλλον, να κάνει ένα στοίχημα για το μέλλον και να θα στοιχηματίσετε στη βελτίωση του ντίζελ ή των ηλεκτροκινητήρων. Εγώ ποτέ δεν θα δώσω μια τέτοια συμβουλή για επενδύσεις. Για ιστορικούς λόγους, επειδή δούλευα στην επιχείρηση, μπορεί να έχω μετοχές στην Daimler Benz και στην BMW. Είχα, τα έχω κρατήσει αυτά για μια δεκαετία και συνεχίζω να τα κρατώ. Νομίζω ότι είναι καλές επιχειρήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι εκεί που δεν έχω επενδύσεις δεν είναι καλές. Πάντως τα πράγματα δεν εξελίσσονται τόσο γρήγορα στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Είπα το δεινόσαυρη ε, θα έλεγα ε, προκλητικά λιγάκι. Οι καινοτομίε έρχονται από ανθρώπους ε, που έφτιαξαν την Τέσλα ή το Uber. Οι πετρελοκινητήρες θα συνεχίσουν να υπάρχουν, να είναι βιώσιμες λύσεις για τους καταναλωτές, αλλά το κοινό θα πρέπει να προσπαθήσει να ανακτήσει εμπιστοσύνη σε μια σωστή επιλογή γύρω από τις μηχανές αυτές. Αυτός είναι ο κίνδυνος και εκεί ακριβώς ε, το σκάνδαλο ε, Dieselgate μας το κατέστρεψε. Α, λες, α, οδηγείς ένα δίζελ, αυτό σημαίνει ότι οδηγείς ένα βρώμικο αυτοκίνητο. Δεν είναι σωστό αυτό. Μας είπατε επίσης ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν εκφράστηκαν και δεν κατήγγυλαν όλα αυτά τα οποία ήταν γνωστά σε πολύ κόσμο. Αν λοιπόν έχετε την δυνατότητα να παρέμβετε για καθορισμό νέων κανόνων, θα πρέπει κυρίως να βελτιώσετε την προστασία ε, των ανθρώπων αυτών ε, που ε, φέρνουν σε επιφάνεια τις απάτες ή να μειώσετε την εκπομπή των καυσαερίων. Κοιτάξτε αν σας κατάλαβα καλά η μείωση των εκπομπών, η διαχείριση του θέματος των εκπομπών είναι κάτι το οποίο σαν κοινωνία πρέπει να κάνουμε και εσείς σαν εκπρόσωποι μας φίλετε να κάνετε. Αν θέλουμε να είμαστε σωστά ενημερωμένοι για αυτούς που είναι στο εσωτερικό των μεγάλων επιχειρήσεων για σκόπιμες παραβιάσεις του νόμου, πρέπει να τους προστατεύσετε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αλλιώς δεν θα συμβεί. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι σαν τον Έντουάρτ Σνόουντεν οι οποίοι ε, επέτρεψαν στην κοινωνία να κάνει βήματα προς τα εμπρός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπατε και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας, όλοι οι επόμενοι ομιλητές ε, ήδη πήραν το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν είστε σύντομοι. Σύντομες ερωτήσεις, σύντομες απαντήσεις. Παρακαλώ. Σύντομα θα επανέλθω στην ερώτηση που έκανε η κυρία Εύη για τους παράγοντες συμβατότητας ή συμμόρφωσης. Ήσασταν ειλικρινείς σε όλες τις ε, απαντήσεις και στην εξής ερώτηση να κάνετε το ίδιο. 1,5 το 2021 εμείς ε, επιβάλαμε στους, δημόσ, στους δεινόσαυρους όρια που θα τους αναγκάσουμε να γίνουν και να τρέχουν σαν λαγί, ή γίναμε και εμείς δεινόσαυροι σαν κι αυτούς. Όπως είπα, και το RDE και οι παράγοντες σύμμορφωσης ε, είναι ένα καλό παράδειγμα διακανονισμού των πραγμάτων. Υπάρχει περνάμε από μία περίοδο όπου μόνο τα τεστ είχαν ε, κάποια ουσία σε μία περίοδο όπου τα τεστ αυτά αποκτούν μία πραγματική αξία. Και δίνεται χρόνο για να το πετύχει αυτό. Ξέρουμε όμως ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι από μόνο του επαρκές. Τώρα είσαστε επιφορτισμένοι να κάνετε νέες διακανονιστικές προτάσεις που θα αποτρέπουν τις απάτες αυτές στο μέλλον όπως και να προσπαθήσει κανείς να εξαπατήσει. Όχι βάζοντας συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά βάζοντας κάποια ανώτατα όρια τα οποία δεν θα πρέπει να παραβιαστούν η κυρία Τούνουν Χόνσταϊν, ε, Φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίασης. Ε, θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι σύντομη. Αλλά μια και είσαστε σύμβουλος, δεν ε, θα σας ρωτήσω, μια και δεν είσαστε σύμβουλος, δεν θα σας ρωτήσω για τις επενδύσεις, αλλά Όσον αφορά το μέλλον, πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι βασικοί τομεί στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε. Μιλήσατε για την προστασία των ε, whistleblowers. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και όταν μιλάμε για τις ε, απάτες, ε, εδώ και πάρα πολύ καιρό προωθούσαμε τους κινητήρες diesel. Η νομοθεσία λοιπόν προώθησε τον ντίζελ. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό με τρόπο που να μην νιώθει ο κόσμος προδομένος. Μήπως μπορείτε να αναφέρετε κάποια θέματα στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε για να προλάβουμε μελλοντικά σκάνδαλα όπως αυτά που είδαμε να μην πάρουμε λάθος δρόμο και να αποφύγουμε μελλοντικά σκάνδαλα. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια ε, ανώτατη τιμή εκπομπών και να υπάρχει τρόπος το κοινό να παρακολουθεί την κατάσταση και να μπορούν να λάβουν εμπεριστατωμένε αποφάσει ε, κατά τι αγορέ προϊόντων. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει τον τομέα στη συμμόρφωση. Εμένα δεν με απασχολεί τόσο πολύ το ντίζελ ή όχι. Εγώ νομίζω ότι το μέλλον ανήκει στην ηλεκτροκινητικότητα. Σε 5-10 χρόνια θα έχει ευρύ αντίκτυπο, αλλά φαίνεται όλα να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το να ρυθμίσουμε τους διζελοκινητήρες, ε, τους βενζινοκινητήρες, ε, τους κινητήρες αερίου κλπ. Ε, θα πρέπει να υπάρχει η ίδια ρύθμιση. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τους κινητήρες υδρογόνου, για παράδειγμα, εάν αναπτυχθούν. Ο κύριος Γιαρπάντη, όχι δεν θέλει. Ο κύριος Σούλτσε. Επειδή προηγουμένως μακρηγόρησα, θα ρωτήσω κάτι σύντομα. Ε, υπάρχει δυνατότητα να ψάξουμε, να βρείτε ή να μας πείτε πόσο κοστίζει η ανάπτυξη ενδεχομένω μια τέτοια συσκευή ε, εξαπάτησης. Είπατε ότι είναι πάρα πολλή δουλειά και μεγάλο μπελά και μα είπατε επίση ότι ε, μετεξελίσσεται αυτό, συντηρείται και αναβαθμίζεται. Πόσο κοστίζει περίπου μια τέτοια ε, ε εφαρμογή λογισμικού και θα σας πω γιατί. Ε, τώρα δεν το μελετήσαμε με τέτοιους όρους. Ε, υπάρχει δυνατότητα στατιστικές πόσο ε, κοστίζει ένα line of code και ένα faction point. Αυτά είναι τα κριτήρια που μετράνε στο λογισμικό στην ανάπτυξη της εφαρμογής. Αν βλέπαμε όλο το λογισμικό θα μπορούσαμε να ε, υπολογίσουμε πόσο κοστίζει και στην πραγματικότητα επειδή αυτό δεν περνάει από το Διοικητικό Συμβούλιο για να εγκριθεί η απάτη, ε, κάπου το έχουν βάλει σε άλλη δαπάνη, σε άλλο κονδύλι και το έχουν κάπως κουκουλώσει. Δηλαδή δεν είναι επίσημη δαπάνη στην εταιρεία. Ναι, να σας πω γιατί ρωτάω. Γιατί είμαι κι εγώ μηχανικός και δούλευα πολλά χρόνια ε, στην ε, βιομηχανία, στους προμηθευτές για τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και εκεί ακόμα και μια βίδα να αγοράζαμε έπρεπε να τη δικαιολογούμε με τιμολόγια και με παραστατικά. Αυτό είναι βαριά δουλειά, κάποιος πρέπει να το έχει εγκρίνει. Πολλοί κόσμος δούλεψε για να αναπτυχθεί. Πώς έγινε τόσο κρυφά και ποια στιγμή και, και μέχρι ποιο επίπεδο ιεραρχία της εταιρεία είναι γνωστό αυτό. Και θέλω να διαφωνήσω σε ένα σημείο μαζί σας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα κάτι τέτοιο να κρύβεται επειδή κάποιος φοβάται μη χάσει τη δουλειά του, μη χάσει το εισόδημά του. Όταν δουλεύεις σε μια τέτοια ε, εταιρεία μπορείς να βρεις άλλο δουλειά ή μπορείς να το συζητήσεις μυστικά σε ένα τσάτρουμ Δεν είναι δυνατό να το κρατάνε κρυφό τόσα πολλά χρόνια τόσο πολλοί άνθρωποι. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα ε, δημόσια, γιατί το ομολόγησε η Volkswagen, το επίπεδο κάτω του Διοικητικού Συμβουλίου, παραθέτω από δικό τους έγγραφο, το ήξερε. Και ξέρουμε ότι παρετήθηκε διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος και διοικητικά συμβούλια επίσης. Άρα κάποια γνώση είχαν ή θα έπρεπε να είχαν, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορούσαν να κρατήσουν τη θέση τους επειδή τα γνώσαν προσωπικά, αλλά είναι πραγματικά ε, προσωπική ε, ε, γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν κρατιέται μυστικό έτσι ρητά, διότι ε, κάποιος το αποφάσισε και ανατέθηκε να γίνει. Και δεν έψαξε κανείς αν είναι ενώνυμο ή παράνομο. Του είπανε κάποιου κάνε κάτι και το έκανε. Είναι μια γκρίζα ζώνη πραγματικά στις κρίσεις. Και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι πολλοί από εκείνους που σήμερα έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευέ στην Αμερική δεν το έκαναν ε, συνειδητά ε, γνωρίζοντας ότι είναι παράνομο ή λάθος. Αλλά προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα ε, αυτό το τρίκ ε, της δοκιμής. Η κυρία Γοβονταλόν παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μας δείξατε ότι το λεγόμενο reverse engineering στην ουσία υπήρξε μια αντιγραφή των μεθόδων τις οποίες χρησιμοποίησε η Bosch και είπατε ότι αυτό μπορεί να ισχύει και για άλλους παροχείς λογισμικών. Μπορείτε να μας πείτε τι λογισμικά είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για εξαπάτηση. <laughs> Και ε, τι μπορείτε να πείτε ε, για κάποιες άλλες επιχειρήσεις λογισμικού που, για τις οποίες μπορεί να έχουμε υποψίες. Υπάρχουν δύο τομείς εδώ. Ο ένας τομέας είναι αυτός που μας δείχνει το ποιοι έχουν κάνει απάτες σε επίπεδο προβληματικό νομικά. Το ξέρουμε από το αμερικανικό νομικό σύστημα και τη Volkswagen. Γιατί εκεί δέχτηκε η Volkswagen, παραδέχτηκε ότι εξαπάτησε. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει η Volkswagen για την Ευρώπη και το είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, νομίζω, ότι και ε, οργανώθηκε μια ακρόαση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο όπου η Volkswagen αρνήθηκε ότι έχει ένα τέτοιο μηχανισμό εξαπάτησης στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν και άλλες μικρότερες τέτοιες απάτες για τη θερμοκρασία, για το χρόνο μέτρησης, για παραφουσκωμένα λάστιχα έτοιμα να σκάσουν Αυτά όλα επηρεάζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ασιατική βιομηχανία. Αυτές δεν είναι κατεξοχήν μηχανισμοί, μάλλον δεν είναι εξαπάτησης. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ναι σας εξαπάτησα με συγκεκριμένους μηχανισμούς. Είναι θέματα που πρέπει να ειδωθούν διαφορετικά όταν ψάχνουμε τις νομικές επιπτώσεις. Αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα δεν είναι το πώς εξαπατούν οι βιομήχανοι. Το θέμα είναι να μην μπορούν. Επιβάλλει κανείς έμπαση περιπτώσει συνθήκες οι οποίες με φυσική χρήση δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο εξαπάτησης. Εφόσον Όταν βάζεις ε, ένα μετρητή ε, στο, στην εξάτμιση βλέπεις ότι η πίεση είναι διαφορετική από τις υποκανονικές συνθήκες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορείς να μετρήσεις με βεβαιότητα και να δεις ε, ποιες είναι οι πραγματικές εκπομπές. Πρέπει να πάμε σε ένα επίπεδο παραπάνω. Όταν μπαίνουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, ιδιαίτερα σε επίπεδο διακανονιστικό, πρέπει να ανέβετε ένα επίπεδο και να προσπαθήσετε να το απλουστεύσετε για να γίνει πιο αποτελεσματικό. Και τέλος η κυρία Ρέιδα. Κύριε Λάγε, μια εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τι πράγματι συνέβη απαντήσατε με ακρίβεια στις ερωτήσεις μας, εκτός από μία, την οποία παραλείψατε. Γι' αυτό θα την επαναλάβω. Είναι η δεύτερη ερώτηση στο σημείο 6. Πώς μάθατε από ευρωπαϊκό ή άλλο κατασκευαστή αυτοκινήτων για πρώτη φορά την χρήση ε, λογισμικού αναστολής. Το έμαθα πρώτη φορά από τον τύπο όταν η Volkswagen το ομολόγησε. Το είπα και στην εισαγωγή. Αυτό ήταν που με κινητοποίησε εμένα. Διάβασα τον σχολιασμό της διεύθυνσης που έλεγε ότι μα, οι μηχανικοί μας ε, ξαπάτησαν. Ε, και έλεγα, μα δεν είναι δυνατόν, ε, δεν, δεν πρόκειται να το πιστέψει κανείς. ναι, όντως. και από ό,τι γνωρίζω ούτε ο Φέληξ το γνώριζε πριν. Δηλαδή, το δικό σας τομέα δεν το γνώριζαν όλοι ότι γίνονται τέτοια πράγματα. Όχι, εγώ εργάζομαι στο τομέα της πληροφορικής, ασχολούμαι με ε, υπολογιστές, λογισμικό και βάσεις δεδομένων. Ε, ε, ε, συνεργαζόμουν φυσικά με τους συναδέλφους από την άλλη πλευρά, αλλά στην BMW δεν ήταν γνωστό ότι η BMW ή οι άλλοι κατασκευαστές ε, εξαπατούσαν τον κόσμο. Είπατε ότι χρειαζόμαστε προστασία των ε, για τους ε, καταδότες δημοσίου συμφέροντος και έχετε προτάσεις ε, και ο τύπος προσπάθησε κάτι ανάλογο το οποίο δεν επέτυχε. Αυτό που βγαίνει στον τύπο είναι ελάχιστα κομματάκια πληροφόρησης από κάποια επιστολή ή κάτι τέτοιο και γι' αυτό ε, ο τύπος ε, αμέσως ενδιαφέρθηκε όταν ο Φέληξ εξέτασε το λογισμικό. τώρα στις Ηνωμένε Πολιτείε, τώρα στην ε, δικαστική διαδικασία για ε, ε, την κατηγορία X. Γίνεται κάτι ανάλογο. Όλοι περιμένουμε τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. δεν ε, καταφέραμε να κινητοποιήσουμε κάποιον που να ανήκει στον πυρήνα ε, να κάνει αποκαλύψεις. Δεν ξέρω γιατί, πάντως ο τύπος δεν κατάφερε να λάβει αρκετέ πληροφορίες ε, και γι' αυτό λυπάμαι, δεν νομίζω θα καταφέρει ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι είναι πιο εύκολο να πάει κανείς στον τύπο που θα προσπαθήσει να προστατεύσει την πηγή του από το να δώσει πληροφορίες σε μια εξεταστική επιτροπή. Και είδαμε τι έχει κάνει η Βρετανική Εξεταστική Επιτροπή. Είναι χρήσιμο να διαβάσει κανείς τις σχετικές εκθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λάνια. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνουμε την σημερινή μας πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Ε, ξεκινήσαμε 9 η ώρα το πρωί, τώρα είναι περασμένες 6. Πολύ ενδιαφέρουσες ακροάσεις είχαμε, η μία ήταν η δική σας. Και σας ευχαριστώ για τις ε, πολύ χρήσιμες ε, παρατηρήσεις σας και σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε και στον ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, διότι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουμε από τα κράτη-μέλη, αλλά έχουμε και εμείς να παίξουμε σημαντικό ρόλο και όσον αφορά την επιβολή του νόμου και όσον αφορά την ε, μελλοντική νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ πιθανό να έχουμε συμπληρωματικές ε, ερωτήσεις ε, να σας υποβάλουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ όλους που αντέξατε μέχρι το τέλος. Οι πέμπτες είναι πάντα δύσκολες, ε, το γνωρίζω αυτό και εγώ πρέπει να προλάβω τρένο για την Αμβέρσα. Υπάρχουν άλλοι όμως που <laughs> πρέπει να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συνάδελφοι, να σας ενημερώσω ότι η επόμενη μας συνάντηση είναι 20, 21, 27 Ιουνίου και 4 Ιουλίου. Και έχουμε και κάποιε ακόμα συναντήσει ε, τον Ιούλιο. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ακόμα διακοπέ. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.